Ε, για την παρουσίαση της μελέτης αυτή στην Επιτροπή μας και να τους ε, συγχαρώ. Είναι πολύ καλή η δουλειά αυτή που έγινε, ε, με πάρα πολύ καλό τρόπο και πάρα πολύ πλήρης η μελέτη και αντιμετωπίζει τα θέματα και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις, τους φραγμούς και τα εμπόδια και τις δυσκολίες των επιγραμμικών πωλήσεων σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των ε, καταναλωτών, τις τεχνικές ε, πώληση ε, των επιχειρήσεων και πολλά άλλα στοιχεία. Είναι πολύ ωφέλιμο αυτό και για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο για να ξέρουμε πώς έχουν οι επιγραμμικές πωλήσει, τι θέλουν οι καταναλωτές και τι προσφέρουν οι επιχειρήσεις και πώς λειτουργούν. Συνοδεύεται η μελέτη και από συστάσεις και προτάσεις που ταυτίζονται σχεδόν απολύτως με τις ε, απόψεις της ομάδας εργασίας ε, της ομάδας μας που παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο αν δεν απατώμε. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν πολύ καλά και ποιες είναι οι αναγκαίες λύσεις για να ε, λανσάρουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και τους φραγμούς για να υπάρξει μια φυσική ε, ανάπτυξη και εδραίωση της εσωτερικής αγοράς και της ηλεκτρονικής εσωτερικής αγοράς. Μεσοπρόθεσμα δεν πρόκειται να έχουμε ενιαία εσωτερική αγορά αν δεν λειτουργήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, πιστεύω. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να βρούμε ένα μέσο, ένα τρόπο που να ανθίσταται στις ε, αλλαγές και να είναι χρήσιμο εργαλείο και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Εμείς επανειλημμένα έχουμε πει και μάλιστα και σε έγγραφο που έχουμε εγκρίνει στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια πέρσι το Σεπτέμβριο ε, ότι ε, χρειάζεται ένα σήμα εμπορικής εγγύησης. Και το λέει και η μελέτη, ε, το προτείνει ως φόρμουλα να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη ε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το σήμα εμπιστοσύνης, λοιπόν, Trustmark, θα μπορούσε να είναι ο φορέας αυτός που μας χρειάζεται και όχι ένα λογότυπο απλώς χρειαζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε και ένα φορέα υποστήριξης ε, πληροφόρησης τρισδιάστατο που να ενημερώνει ε, για όλους ε, τους ενεχομένους και όλους τους ενδιαφερομένους. Όπως είπα και τον Ιούλιο και επανενέλαβα πρόσφατα, η έξοδος από την κρίση έχει ψηφιακή μορφή και θα πρέπει οπωσδήποτε να ανασκουμποθούμε για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Άκουσα και τον πρόεδρο της Επιτροπής μας και είναι πολύ πιθανό να διατηρηθεί ομάδα εργασία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Λοιπόν, εκεί ίσως θα ήταν ο φυσικός χώρος να γίνεται αυτή η συζήτηση, να παραμείνει ανοιχτή, να ανταλλάσσουμε απόψει με τους ε, συντάκτες αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας ε, μελέτης. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές αύριο για τη μελλοντική εντολή. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Άγκστρομ. Ο κ. Άγκστρομ θέλει το λόγο και του τον δίνω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την πώληση ψηφιακή νομικών αγαθών. Στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είχαμε μία ομάδα εργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία συνέρχεται ανά το χρόνο με εμπειρογνώμονες και φτάσαμε στο ίδιο συμπέρασμα με αυτή τη μελέτη όταν μιλάμε για ψηφιακό περιεχόμενο. Είναι δυνατόν να ανταγωνιστούμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι στη, στη Σουηδία μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το περιεχόμενο με κατέβασμα στοιχείων, δηλαδή με αυτό το downloading. Αυτά είναι πολύ καλά νέα, αν θέλουμε νομικές εναλλακτικές λύσεις. Όμως δεν υπάρχει πανευρωπαϊκό περιεχόμενο, πανευρωπαϊκές προσφορές. γιατί στην ομάδα εργασία μας θα ήθελα να πω ότι σε επίπεδο 27 θα έπρεπε να υποβάλουμε συγκεκριμένες προσφορές γιατί σε κάθε χώρα θα πρέπει να γίνουν ε, διαπραγματεύσεις με αρκετούς ε, διαπραγματευτές και αυτό δεν είναι εφικτό και επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια όταν μιλάμε για συλλογή στοιχείων, σε κάθε χώρα ερχόμαστε σε διαπραγματεύσεις με τις επιχειρήσεις προσφορών και όταν συλλέξουμε τα στοιχεία βλέπουμε ότι φτάνουμε στο 100% αλλά δεν υπάρχει διαφανής διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πρόβλημα, δηλαδή ο κατακαιρματισμός των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι πρέπει να κάνει σε αυτό τον τομέα, διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα. Έχω την εντύπωση όμως ότι τίποτα δεν θα προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ένας ενιαίος τίτλος πνευματικών δικαιωμάτων και οι προτάσεις διαφάνειας στις ε, επιχειρήσης προσφορών δεν φτάνει σε κάτι συγκεκριμένο. Από πλευράς Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων φτάσαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σε σχέση με την ψηφιακή αγορά. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει κάτι έτσι ώστε να αντιταχθούμε στους ε, μεγάλους φορείς οι οποίοι δεν θέλουν αλλαγές. Θέλουν να υπάρξει στασιμότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αντιταχθεί σε αυτό. Διαφορετικά θα είμαστε στην ίδια κατάσταση με τη σημερινή. Και το Pirate Bay θα είναι ο μόνος μεγάλος πάροχος. Αυτά είναι τα σχόλια. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη συνεισφορά. Θα το συζητήσουμε και στους συντονιστές, διότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θέλει να απαντήσει στο έγγραφο της Επιτροπής για τα πνευματικά δικαιώματα. Γι' αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταπαντήσουμε θα πρέπει όλα να τα εντάξουμε σε ε, ένα συγκεκριμένο, στα συμφραζόμενα υπάρχουν. Η κυρία Λαμόν νομίζω ότι θα ήθελε να απαντήσει από την Κομισιόν και νομίζω ότι θα έχετε και ένα αντίγραφο αυτού του, αυτό των δεδομένων. Κομισιόν, κυρία Λαμόν. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τα πνευματικά δικαιώματα ιδιαίτερα, αλλά να εντάξω αυτές τις εργασίες στα συμφραζόμενα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η έρευνα αυτή φτάνει εγκαίρως, διότι αυτή τη στιγμή Μιλάμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα προβούμε σε μία μελέτη για τις μηχανές αναζήτησης και όλα τα σχετικά και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπεται να εισαχθεί στο παράρτημα του εγγράφου. Η ανακοίνωσή μας θα έχει πολιτικό περιεχόμενο και προσπαθούμε να ορίσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση έτσι ώστε να άρουμε τα προσκόμματα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μπορώ λοιπόν να πω ότι όλα τα θέματα που εφήγησαν στην ομάδα εργασίας και σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται έτσι ώστε να επιλύσουμε διαφορές, να δούμε τι θα, γίνουμε, τι θα γίνει με τις παραδόσεις, ε, τις πληρωμές, την προστασία δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο και ούτω καθεξής. Δηλαδή να ορίσουμε τους επιμέρους όρους και να προβάλλουμε και ένα πρόγραμμα δράσης για την άρση των εμποδίων. Ελπίζουμε πριν από το τέλος του έτους να σας υποβάλουμε αυτό το έγγραφο έτσι ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευπρόσδεκτη η πρόταση και μπορείτε να λάβετε και ένα αντίτυπο της μελέτης. Μίλλερ και Νταμγκάρτ θέλετε να προβείτε σε σχόλια πριν κλείσουμε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας πω ότι η ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να βρούμε έναν διάβλο μεταφοράς, διάβλο διάδοσης, έτσι ώστε να μην είναι τόσο κατακερματισμένος όπως μέχρι τώρα. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη δράση εξέβρεσης διάβλων. Ε, συμφωνούμε, λέει ο Πρόεδρος, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να προβάλλουμε κατευθυντήριες γραμμές. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και οι πολίτες αναμένουν πολλά από εμάς, αναμένουν βοήθεια από εμάς και γι' αυτό θα πρέπει να προβάλλουμε προτάσεις ζωτικής σημασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θα το δούμε το θέμα με τον κύριο Αρίας και με την ομάδα εργασίας και θα λάβουμε αποφάσεις για την πολιτική αυτή. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με, το πρώτο, με την πρώτη μεγάλη έκθεση που μας απασχολεί. Πρόκειται για την έκθεση McClarkin είναι μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για έναν τομέα που μας ε, ενδιαφέρει εδώ και μακρύ χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει και μία πράσινη βίβλο, έτσι ώστε να ορίσουμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Η κυρία Μακλάρκιν, λοιπόν, θα μας παρουσιάσει αυτό το έγγραφο και μετά θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις που είναι παρόντες. Η κυρία Λεγκρίπ δεν είναι εδώ. Εξ ονόματος ε, του ΕΛΚΟ, κύριο Σβάμπη. Ίσως, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος άλλος θα λάβει το λόγο. Η κυρία Βανιού είναι εδώ. Μπουζόη, ο κύριος Μπουζόη δεν είναι εδώ. Θα δούμε ποιοι είναι. Τούρενεν επίσης, η κυρία Τούρενεν είναι εδώ. Καλημέρα σας. Η κυρία Σβένσον δεν είναι ε, εδώ διότι έπρεπε να ε, παραιτηθεί από το Κοινοβούλιο. Και Υπάρχει και, έχουμε και την Κομισιόν, όλη την ομάδα, η οποία είναι παρούσα. Δίνω το λόγο στην κυρία Μακλάρκιν για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας καλημερίζω όλους. Ελπίζω να περάσατε ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθώ διότι ε, είναι δύσκολη η αρχή. Όπως ξέρετε, η έκθεση αυτή είχε συνταχθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να ρίξατε μία ματιά. Βασιζόμαστε σε διάφορα έγγραφα της Επιτροπής που είχαμε πριν από την καλοκαιρινή διακοπή σε σχέση με την αξιολόγηση και την πράσινη βίβλο. Όπως ξέρετε είχαμε έναν διάλογο με την Κομισιόν σε επιμέρους θέματα και σας ευχαριστώ πολύ. Οι σκιώδεις μας βοήθησαν ιδιαίτερα με σκέψεις στα πρώιμα στάδια αυτής της έκθεσης και θα ήθελα να λάβουμε υπόψη όλες τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων Ελπίζω αυτή η οδηγία να είναι πιο αποδοτική για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Προσπαθούμε να έχουμε ένα πραγματικό input για τις προτάσεις της Επιτροπής αργότερα. Ήρθα σε επαφή με πολλά επαγγέλματα και επαγγελματικούς φορείς και μιλάμε για βασικές υπηρεσίες ανά την Ευρωπαϊκή ε- Ένωση και ποιοτικά στοιχεία στην ενιαία αγορά. Θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο θέλουν να, υπάρχει, ε, ε, να υπάρχουν σωστοί διάβλοι λειτουργία των συστημάτων και ποιοτικέ υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά ποιοτικά συστήματα και να μην έχουμε διοικητικά προσκόμματα. Πολλοί επαγγελματίες και ρυθμιστές, καθώς και οι Κομισιόν, είπαν ότι η αμοιβαία αναγνώριση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να απλουστευτεί, διότι υπάρχουν απαρχαιωμένα στοιχεία, έχουμε ε, νέες τεχνολογίες, τις οποίες δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και πολλά στοιχεία έχουν ξεπεραστεί στον 21ο αιώνα οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν σε πραγματική απασχόληση έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε ενεργητικό ρόλο στην ενιαία αγορά. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες ρυθμίσεις στον τομέα της υγείας έφνης, έτσι ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην οδηγία του 2005 για να μπορέσουμε να έχουμε ευέλικτες ε, αγορές εργασίες και να έχουμε καλύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε όλα τα κράτη-μέλη και να έχουμε υψηλές υπηρεσίες για τους καταναλωτές και τους ασθενείς. Μετά από δημόσια διαβούλευση βλέπουμε ότι η οδηγία φτάνει σε, αυτούς, φτάνει αυτά τα αποτελέσματα, λαμβάνει υπόψη πραγματιστικά στοιχεία και υπάρχει αναγνώριση ανατομής για να επιταχύνουμε τη διαδικασία αναγνώρισης. Υπάρχουν όμως το μίσο που θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές και θα ήθελα να δούμε λεπτομεριακά. Ήταν πολύ κοπιώδης αυτή η διαδικασία έτσι ώστε να ρυθμίσουμε διάφορα επαγγέλματα και επίσης πολλά κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να μεταφέρουν αυτή την οδηγία το Solvit και άλλοι φορείς είδαν ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση και μόνο σε ένα 20% μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχουν πολλά παράπονα και προσφυγές διότι δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα και πολλές φορές δεν ξέρουν οι επαγγελματικοί φορείς τι έγγραφα πρέπει να υποβάλουν για την πλήρη αναγνώριση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση από την παρούσα κατάσταση. Δεν υπάρχει ε, ευρεία εμπιστοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη έτσι ώστε οι διατάξεις να είναι απλές και πιο αποτελεσματικές και να λειτουργούν τάχιστα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε contact points σημεία επαφής έτσι ώστε να προωθήσουμε τον διάλογο μεταξύ αρμοδίων αρχών η πράσινη βίβλος της Επιτροπής προβάλλει σημαντικά στοιχεία, ιδιαίτερα για την πρόσβαση online, για να ξέρουν οι φορείς ποια έγγραφα χρειάζονται και με ποιες αρχές θα πρέπει να έρθουν σε επαφή. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μία online διαδικασία υποβολής εγγράφων για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης όμως θα πρέπει να ε, παγιοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες με, βάλει, με βάση συγκεκριμένες πύλες, διαδικτυακές πύλες, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να υποβάλει τα στοιχεία σε συγκεκριμένες πύλες. Στην οδηγία του 2005 υπάρχουν διατάξεις που θα πρέπει να αλλάξουν, διότι αφορούν μια κατάσταση που ίσχυε 30 χρόνια πριν. Όμως στο, στην Πράσινη Βίβλο η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατεξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει κατάρτισης έτσι ώστε να υπάρχει και καλή εποπτεία για τις αποφάσεις. Επίσης, συγκεκριμένοι τομείς της οδηγίας μας απασχόλησαν. Θα πρέπει να υπάρχει μια επαγγελματική κάρτα, όπως ορίζεται στην Πράσινη Βίβλο με πιλωτικές έρευνες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επαγγελματική κάρτα θα επιταχύνει τη διαδικασία αναγνώρισης έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Τα αποτελέσματα των πιλωτικών μελετών θα υποβληθούν αργότερα στο έτος. Όμως η δημόσια διαζή θα πρέπει να προωθηθεί σε σχέση με το κόστος και την αξιοποίηση και το βάσιμο αυτό των δεδομένων. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποια προστιθέμενη αξία μας δίνει πραγματικά η επαγγελματική κάρτα. Θεωρούμε ότι αυτή η κάρτα θα πρέπει να ακολουθεί μια ε, εθελούσια βάση, να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και να ε, βοηθά τους ρυθμιστές ως προς την εφαρμογή. Γι' αυτό αυτή η εκούσια κάρτα θα πρέπει να βασίζεται στο, σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα όπως το IMI. Το IMI θεωρείται ε, αποτελεσματικό μέσο για τις πληροφορίες αυτές θα πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε το IMI έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν σωστά. Επίσης θα πρέπει να δούμε πού δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή έτσι ώστε να έχουμε συμμετοχή των αρμοδίων αρχών για να βοηθήσουμε τα επαγγέλματα και η οδηγία επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να προβάλλει μία αρχή προειδοποίησης και θα πρέπει να διευρύνουμε το IMI σε ένα σύστημα προειδοποίησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Επίσης, η μερική πρόσβαση είναι ένα άλλο μέσο για να βοηθήσουμε την κινητικότητα. Η διαβούλευση δείχνει ότι οι αρμόδιες αρχές, οι επαγγελματικοί φορείς θέλουν να ε, διευρυνθεί και να, αλλάξει, να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα έμπρακτα. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρης αξιολόγηση και να δούμε και ιδιαίτερα τον τομέα της υγείας και ασφάλειας. Επίσης χρειάζονται μέσα, μέτρα αντιστάθμισης έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να είναι σίγουρες ότι υπάρχουν σωστά προσόντα και μέσα. Υπάρχουν όμως περιστάσεις ώστε ε, να χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα όχι αναλογικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν και μέτρα αντιστάθμισης και τα μέσα αυτά να είναι διαφανή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις αλλαγές που επέρχονται γιατί πολλές φορές οι νέοι αντιμετωπίζουν πολλά προσκόμματα για την ελεύθερη ε, διακίνηση και την αναγνώριση των προσόντων τους. Δηλαδή δεν μπορούν να ε, ασκήσουν το επάγγελμά τους ε, γιατί υπάρχουν προσκόμματα ως προς και την υπηκότητα. Η διαδικασία της Μπολόνιας είναι πολύ σημαντική και η ΙΜΚΟ θα αποφανθεί τις επερχόμενες εβδομάδες. Η Πράσινη Βίβλος όμως θεωρεί ότι θα πρέπει να ε, δεχτούμε και τα δεδομένα από τις τρίτες χώρες. Όμως, επειδή το παρόν σύστημα είναι περίπλοκο, νομίζω ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες χώρες, διότι αυτό θα φόρτωνε ιδιαίτερα το σύστημα. Επίσης, ως προς την προσωρινή κινητικότητα, η οδηγία του 2005 εισάγει νέα στοιχεία έτσι ώστε να έχουμε υπηρεσίες βραχυπρόθεσμα με βάση τις επιλογές των καταναλωτών και οι επαγγελματίες να μπορούν να εργάζονται σε άλλα κράτη-μέλη χωρίς να υπάρχουν περίπλοκα συστήματα. Όμως θεωρούμε ότι η προσωρινή ε, κινητικότητα θα οδηγούσε σε forum shopping και δεν θα βοηθούσαμε στην καλή προσέγγιση. Άρα η οδηγία κατέστησε δύσκολο ε, τον ε, χρονικό προσδιορισμό. Γι' αυτό θα ήθελα το άρθρο 7 να διασαφινιστεί από, τον, από την Κομισιόν η κινητικότητα είναι πολύ σημαντική, είτε είναι προσωρινή είτε μόνιμη. Αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο επαπειλείται η δημόσια υγεία και ασφάλεια. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο γλωσσικό. Έγινε μια πολύ ζωηρή συζήτηση έτσι ώστε οι επαγγελματίες να έχουν τα γλωσσικά προσόντα για να μπορέσουν να εργαστούν σε ένα άλλο κράτος μέλος, ιδιαίτερα στον τομέα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Δεν υπάρχουν επαρκείς διασαφήσεις για τα, για τα μέσα που θα μπορούσαν να προβληθούν η Κομισιόν μιλά για μία αναπερίπτωση προσέγγισης στα θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Αυτό όμως θα πρέπει να διασαφινιστεί σε σχέση με τον κώδικα συμπεριφοράς και να εισαγάγουμε νέα στοιχεία αναγνώρισης γλωσσικών προσόντων. Θα πρέπει να υπάρχει αναλογική προσέγγιση και να μην αποτελέσει πρόσκομα στην κινητικότητα. Προσπάθησα να δω κάθε πτυχή της οδηγίας. Η Κομισιόν ασχολήθηκε ευρέως με αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο. Βλέπουμε ότι για πολλούς επαγγελματίες λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα, όμως η αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί και πολλές φορές χρειάζεται εξυγχρονισμός. Η επαγγελματική κάρτα και άλλα μέτρα θα πρέπει να αξιολογηθούν πριν εφαρμοστούν. Θα πρέπει να δούμε και τα γλωσσικά προσόντα και να προσπαθούμε προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τον τομέα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να επιταχύνουμε το σύστημα αμοιβαία αναγνώρισης, ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελματίες, έτσι ώστε να υπάρχει δίκαιη προσέγγιση. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, στις 22 Σεπτεμβρίου έχουμε, την, έχουμε ορίσει την προθεσμία και στις 19 θα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη η οποία θα είναι ενδιαφέρουσα για την υποφαινόμενη και τους άλλους ε, σκιώδεις. Στις 17 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε και το Νοέμβριο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Ελπίζω να στάθηκε χρήσιμη αυτή η παρουσίαση και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Την κυρία Μακάκη είναι πάρα πολύ σαφής η παρουσίαση και πολύ καλά δομημένη και θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Τώρα θα παρακαλέσω τους και ηγητές να μας δώσουν τις απόψεις τους. Και αν θέλουν και άλλοι ε, συνάδελφοι, παρακαλώ να ζητήσουν το λόγο. Κορόντε Κάμπο Σουβά και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ προς το παρόν. Και η κυρία Κουτιέρες. Καλώ ορίσατε. Νομίζω εκπροσωπείτε την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, εδώ. Είστε σχεδόν η γνωμοδότηση. Και ε, άλλοι συνάδελφοι αργότερα. σας έγραφε στον κατάλογο. Μάλιστα. Α, και ο κύριος Φάπα, παλίμονο. Η κυρία Λεγκρίπ και θα δούμε με τη σειρά. Ο κύριος Μπουζό ήρθε. Πρώτα η κυρία Λεγκρίπ όμως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά ξαναβρίσκω τα μέλη της Επιτροπής μας της Εσωτερικής Αγοράς, υπ' ευκαιρία της ε, επανόδου μας, ιδιαίτερα για τόσο σημαντικό θέμα που είναι το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, μπορούμε να συνεχίσουμε την αλλαγή απόψεων ε, που είχαμε αρχίσει πριν τις θερινές διακοπές η αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων είναι βασικότατο στοιχείο, ένα από τα 12 που είχε εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε τονίσει ο Επίτροπος Μπαρνιέ ως ε, εκ των για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. αυτό το θέμα μας απασχολεί σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο θα απασχολήσει και την Επιτροπή μας αλλά και το Κοινοβούλιο επί σειρά μηνών. Ευχαριστώ την κυρία Μακλάρκιν για το σχέδιο έκθεσης που σήμερα μας υποβάλλει. Όπως είπε και η ίδια είναι καρπός ε, πρώτερης συνεννόησης και συνεργασίας ε, με τους σκιώδεις συγητές. Έδειξε μεγάλη προθυμία και μεγάλο πνεύμα ε, συνένεσης και επικοδομητικό η συγγήτρια και δεν μας εκπλήσει ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με το σχέδιο έκθεσής της. Η ομάδα μου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, επανειλημμένα έχει τονίσει αυτά τα θέματα και εγώ προσωπικά είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω σε προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση, καμία διαφωνία στα μεγάλα θέματα και αυτό είναι χαρά για και και συγητή κάθε φορά. Ε, Επί τη βάση της έκθεσης της συναδέλφου και βασιζόμενοι όμως στα τέσσερα κεφάλαια στα οποία ε, έχει χτίσει την έκθεσή της, έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, απλοποίηση λέει των διαδικασιών για τους πολίτες. Βεβαίως είναι προς όφελος των πολιτών και είναι μέγας στόχος. Ξέρουμε σε πόσο και σε ποιο βαθμό η γραφειοκρατία ή η ολιγορία των διαδικασιών είναι απαράδεκτη και αφόρητη για πολλούς ε, πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και τεχνολογίας. Βεβαίως, θα πρέπει να υπάρξει μια ηλεκτρονική πύλη ε, για να ενημερώνει ε, έγκυρα και έγκαιρα τους πολίτες. Βεβαίως και όλες οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν ε, αυτή την δικτυακή πύλη. Συνεχίζω πάντα για την απλούστευση ή την απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντελώς απαραίτητο να ε, έχουμε ε, πιο εναρμονισμένες ή με καλύτερα συντονισμένες απαιτήσει αρχικές. Δηλαδή στην εκπαίδευση εννοώ, να συντονίζονται καλύτερα οι αρμόδιες αρχές από τα κράτη-μέλη εκ των προτέρων και στις δραστηριότητες, στις επαγγελματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στα επαγγέλματα υγείας έχουμε συμφέρον να δούμε ε, ποια είναι η εκάστοτε επαγγελματική πραγματικότητα ε, από χώρα σε χώρα. Γιατί διαπιστώνουμε ότι μπορεί να είναι μεγάλες οι αποκλήσεις και στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και στον τρόπο άσκησης ε, του επαγγέλματος αυτού. Επίσης, Ε, θα πρέπει να εναρμονιστεί καλύτερα το θέμα των αποδεικτικών στοιχείων της επαγγελματικής πείρας. Και εδώ χρειάζεται απλοποίηση. Δηλαδή, πώς θα πιστοποιείται η επαγγελματική πείρα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αρμόδιος εθνικός φορέας ή ένας οργανισμός, σε βάση περιπτώσει, που θα έχει επιφορτιστεί στη χώρα προέλευσης ε, για να πιστοποιεί την πείρα του επαγγελματία. Και ε, τελειώνω για το πρώτο κεφάλαιο, βεβαίως. Είχα την ευκαιρία να το πω και σε προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων ο αριθμός των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται είναι από 4.600 4.700. Εν πάση περιπτώσει, είτε το ένα νούμερο ισχύει είτε το άλλο, είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων αυτός. Θα πρέπει κάπως να το συντονίσουμε και να μειώσουμε τον αριθμό των επαγγελμάτων. Το δεύτερο κεφάλαιο επιγράφεται ενημέρωση ή επικαιροποίηση των υφισταμένων διατάξεων. Βεβαίως χρειάζεται καλύτερη ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τα συστήματα υγεία, Λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βεβαίω όλα αυτά περιγράφονται λεπτομερώ στην έκθεση Μακλάρκιν και συμφωνώ και προσυπογράφω. Κεφάλαιο τρίτον. Αναβάθμιση λέει της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Εδώ θίγει ένα θέμα πάρα πολύ ακαθόδες και λεπτό, τουλάχιστον για τους πολίτες, που είναι το μέσο της υγείας. Και έχουν ειδικό καθεστώς τα επαγγέλματα υγείας και επαγγελματίες γιατί είναι ε, ξεχωριστές και οι απαιτήσει και οι ιδιαιτερότητες. Ε, έχουμε συναντήσει όλοι μας επαγγελματίες υγείας, είναι ιδιαίτερος ο κλάδος και οι απαιτήσει, επαναλαμβάνω, ορισμένοι μάλιστα εκφράζουν ε, το πόθο το όνειρο να υπάρξει ad hoc οδηγία ξεχωριστή αφιερωμένη στα επαγγέλματα υγεία. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, ε, δεν θέλουμε τόσο πολύ να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο, αλλά να ε, επιμείνουμε ότι έχει ίδιε απαιτήσει αυτό ο κλάδο και ιδιαιτερότητε. Και ακριβώ εκεί πώς να το πω, θα πρέπει καλύτερα να ταυτοποιήσουμε τις δραστηριότητες και να γνωρίζουμε τις επαγγελματικέ δραστηριότητες ε, των επαγγελμάτων υγείας, γιατί τίθεται το θέμα των ε, προσόντων της επαγγελματική κατάρτισης. Αλλά καλό θα ήταν, πέρα από τα προγράμματα σπουδών, ας πούμε, εκ των προτέρων, και το ξέρω ότι δεν υπάρχει ακόμα σε επίπεδο 27 αυτό, να έχουμε ένα πίνακα όσο γίνεται πιο εξαντλητικό των ιατρικών δραστηριοτήτων και των διαφορών που έχουμε από χώρα σε χώρα. Όταν αναφερόμαστε σε κάποια ειδικότητα ή σε κάποια δραστηριότητα ενός επαγγέλματος υγείας. Υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο γνωστικό που θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε. Και η μερική πρόσβαση επίσης είναι ένα θέμα καθόδες. Τι θα πει, η μερική πρόσβαση είναι δύσκολο να ενδεχθεί στην πράξη. Και εκεί υπάρχουν επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί και τις έχουμε ακούσει κι εμείς. Επίσης ε, και τα προσόντα που αποκτώνται σε τρίτες χώρες. Πώς θα γίνεται η αναγνώριση και η πιστοποίηση αυτών. Euh, και ε, ανησυχούν πραγματικά οι επαγγελματίες. Και βεβαίως το θέμα των γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων, ε, όλοι οι επαγγελματίες που ε, συναντήσαμε τονίζουν ε, τις βαθιές τους ανησυχίες από αυτού και ζητούν να βελτιωθεί η κατάσταση και να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη αυτό το θέμα των γλωσσικών δεξιοτήτων. Αλλά η έκθεση Μακλάρκιν είναι σαφέστατη από αυτού και συμφωνώ απολύτως. Τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, ενσωμάτωση των επαγγελματιών και ενστάλλαξη εμπιστοσύνης, λέει, στο σύστημα. Η ενσωμάτωση των επαγγελματιών, η ένταξή τους είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης. Ε, μας ζητούν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι από όλα τα επαγγέλματα να είναι όσο γίνεται περισσότερο ενταγμένοι στα συστήματα, με τις επαγγελματικές τους ενώσεις, με τους συλλόγους, με τις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στις χώρες τους, όσο γίνεται να ενέχονται σε αυτό το σύστημα, να είναι ενταγμένοι και ενσωματωμένοι ε, στα συστήματα αναγνώρισης. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το σύστημα ΙΜΗ αυτό, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί, να επεκταθεί, ε, συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια. Ε, μηχανισμός ε, προειδοποίησης και βέβαια ε, το ζητούν οπωσδήποτε οι επαγγελματίες, αρχής γενομένης από τους επαγγελματίες υγείας, χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και τέλος η επαγγελματική κάρτα, τι είναι αυτό, είναι προβληματικό. Και γεννάει βέβαια και πολλές ελπίδες. Γίνονται διάφορες πιλωτικές προσεγγίσεις και πολλοί επαγγελματίες έχουν ε, εργαστεί και πολλά επαγγέλματα είναι ήδη έτοιμα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ερωτηματικά ως προς το τεχνικό σκέλος, το οικονομικό, ε, το νομικό, γιατί η προστασία και ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε Ω προτεραιότητα στο Κοινοβούλιο και μια τέτοια επαγγελματική κάρτα θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε προαιρετική, έτσι κι αλλιώ, δεν ε, πρόκειται να επιβάλλουμε οτιδήποτε σε επαγγέλματα που δεν το ζητούν ή μάλιστα ε, χειρότερο θα το θεωρούν ως απειλή ή ε, διακύβευση της ασφάλειάς τους. Αλλά για την εσωτερική αγορά αλλά και για την Ευρώπη των πολιτών, την οποία όλοι προσδοκούμε, χρειάζεται και κάποια προσέγγιση έτσι πιο ενεργή, πιο θελησιοκρατική. Να πούμε ότι θέλουμε ε, να υπάρχει επαγγελματική κάρτα, αλλά πάντα προαιρετική. Πάντως να γίνει κάτι συγκεκριμένο, απτό, χειροπιαστό, στην κυριολεξία Και αυτό δείχνει ε, ισχυρή πολιτική βούληση και στένος από την πλευρά των βουλευτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρώπη των πολιτών. Αυτά. Λοιπόν, μπορούμε να βασιστούμε στην εμπειρία που ήδη έχουν πολύ επαγγελματική κλάδοι και να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι και θέλουμε και μπορούμε για την επαγγελματική κάρτα, επαναλαμβάνω, είναι προαιρετική. Αυτά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω να ακούσω, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα έχουν να πούν οι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι σκιώδεις ηγητές. Ευχαριστώ την κυρία να έχει κάνει πάρα πολύ εμπειριαστατωμένη δουλειά ε, και με μεγάλο επικοδομητικό πνεύμα και συνεννόηση. Και... Είμαι βέβαια ότι και κατά τη ε, διάρκεια τη σύνταξη των τροπολογιών θα συνεχιστεί αυτή η στάση τη ηγητρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεκρύπ. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας ε, είπατε και προτείνατε και στην έκθεση κυρίας Μακλάρκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, ευχηθώ καλή επιστροφή ε, μέσα στα πλαίσια αυτού αυτό των κακών καιρικών συνθήκων, γκρίζος ο ουρανός. Σε πάση περιπτώσει θα πρέπει να φτάσουμε σε μία συνένεση και εμείς θα πρέπει να μετατρέψουμε αυτόν τον γκρίζο ουρανό σε γαλάζιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακλάρκιν και εγώ, όπως και η κυρία Λεγκρίπ, θα ήθελα να είμαι σύντομη, διότι πολλοί έχουν πολλά να πούν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, μία ευρύτατη προσέγγιση και πολύ, οι περισσότεροι δεχόμαστε το περιεχόμενο. Θα ήθελα να το δούμε ανακεφάλαιο και θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια επί του θέματος που είναι ένα θέμα κλειδί για την Ευρώπη των πολιτών και των επαγγελματιών, που είναι όλοι πολίτες. Στο πρώτο μέρος Μιλήσατε για προσωρινή παροχή υπηρεσιών. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα κλειδί και νομίζω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα πρέπει να τονίσουμε τι επιθυμούμε, διότι δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε την ε, προηγούμενη δήλωση και ανακοίνωση της Κομισιό. Η παράγραφος 5, ε, 5 θα πρέπει να αναφέρεται στον ε, κώδικα συμπεριφοράς, θα πρέπει να δούμε τι επιθυμούμε. Στη δεύτερη παράγραφο φύγεται ένα άλλο θέμα που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και όπως ορίζει και η Πράσινη Βιβλός, νομίζω όταν μιλάμε για διαρκή κατάρτιση θα πρέπει να μιλάμε για ελάχιστες προαπαιτήσεις. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ορίσουμε την αναγκαιότητα και μιας γλωσσικής καθαρά κατάρτισης ενός κοινού πλαισίου και να πούμε τι επιθυμούμε σε σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνιας να ορίσουμε ορισμένα σημεία της διαδικασίας της Μπολόνιας και να δούμε ποιες είναι και οι δυσκολίες που δημιουργεί αυτή η διαδικασία της Μπολόνιας και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέραν αυτής. Στα πλαίσια του τρίτου κεφαλαίου θίξατε το θέμα της μερικής ε, πρόσβασης. Η κυρία Λεγκρίπ μας είπε τι σκέφτεται και συμμερίζομαι αυτά που είπε. Νομίζω όμως θα πρέπει να προσέξουμε να μην περιορίσουμε αυτή την αρχή της ε, προσωρινής πρόσβασης στον τομέα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Θα πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για ασφάλεια. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και νομίζω ότι αυτό το θέμα της μερικής πρόσβασης θα πρέπει να αφορά μια γενικότερη συλλογιστική που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το εντάξουμε αλλού. Για να μην επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Λεγκρίπ, θα ήθελα να σταθώ στην επαγγελματική κάρτα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η επαγγελματική αυτή κάρτα ε, εμπεριέχει ένα κόστος. Θα πρέπει να δούμε, να κάνουμε μία ανάλυση κόστους ωφέλειας και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες αυτής της κάρτας με βάση την ε, προηγούμενη πείρα μας. Συμμερίζομαι αυτά που είπε η κυρία Λεγκρίπ Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να δούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη πολλοί πολίτες αμφιβάλλουν έχουν εκφράσει αμφιβολίες ως προς το ευρωπαϊκό σχέδιο και προγραμματισμό. Παλινοδούμε δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία νέα εμπιστοσύνη προς τους πολίτες, είτε είναι χρήστες, πελάτες, ασθενείς, επαγγελματίες. Θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη φιλοδοξία για να προετοιμάσουμε το μέλλον των νέων. Αυτό το προανέφεραν και η κυρία Λεγκρίπ και η κυρία Μακλάρκιν, γιατί μαζί τους ε, θα οικοδομήσουμε ένα νέο μέλλον σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Θα πρέπει τουλάχιστον να τους δώσουμε τα μέσα για να μπορέσουν να το κάνουν. Και αυτή η επαγγελματική κάρτα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Είναι ένα αναγκαίο μέσο για αυτή την Ευρώπη των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ <clears throat> κύριε Βερνιό για την παρέμβασή σας καθώς και για την αισιοδοξία που διέκρινε τα λόγια σας. Ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μακλάρκιν για την ε, σκληρή δουλειά που έκανε. Η έκθεσή, μας, η έκθεσή της μάλλον είναι καλά διαρθρωμένη και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία για την βελτίωση των κανόνων αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Εγώ συμφωνώ με ορισμένα πράγματα. Ιδίω μου αρέσει η ιδέα της χρήσης της βελτίωσης της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας της επικοινωνίας για την πρόσβαση στους πολίτες. Εδώ χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, διότι μου φαίνεται λίγο δύσκολο να συνδυαστούν το Solvit, οι εθνικές αρχές και οι διεθνείς αρχές όλες μαζί. Εδώ με κάποιο τρόπο πρέπει να συντονίζεται η συνεργασία αυτή από κάποιον. Επίσης, είναι σωστό που διευκρινίζεται η ιδέα της προσωρινής κινητικότητας. Εδώ προσθέτω ότι η προσωρινή κινητικότητα ίσως διευκολυνθεί εάν καταστεί δυνατόν να στέλνεται η σχετική δήλωση μέσω email. Από την άλλη μεριά, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, θεωρώ ότι η δήλωση πρέπει να έχει ε, ισχύ σε όλη τη χώρα. Γιατί ε, αλλιώς θα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα. Μέτρα αντιστάθμισης είναι σημαντικά για την προστασία των ε, ασθενών και καταναλωτών. Νομίζω ότι για να αποφύγουμε τα αρνητικά θα πρέπει να έχουμε συνολικές ε, κατευθύνες γραμμές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρήση των δυνατοτήτων αυτών που θα οδηγήσουν και σε πιο ε, ομοιόμορφες πρακτικές. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές παρά ένας κώδικας διοντολογίας που ίσως είναι παραπλανητικός. Ασφαλώς και χρειάζεται υψηλός βαθμός εναρμόνισης, αυτός θα ήταν ιδεώδης μάλλον. Αν και αν ακόμα υπάρξουν ε, ευρωπαϊκά ε, ε, συνολικά προγράμματα, νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό και γι' αυτό προτείνω να γίνει προσπάθεια να λειτουργήσουν οι κοινέ πλατφόρμες. Για τις απαιτήσει τώρα σχετικά με τα αυτόματα συστήματα αναγνώρισης θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι διατυπώσεις ώστε να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για τις ελάχιστες προδιαγραφές ώστε έτσι, έτσι ώστε να συντονιστούν με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και βεβαίως να αναθεωρούνται αυτές σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ επίσης για την προσοχή που δόθηκε στην προστασία των ασθενών και κυρίως για την ενημέρωση όταν έχει επιβληθεί κάποια κύρωση σε έναν επαγγελματία και όταν δεν, δεν καλύπτεται η περίπτωσή του από τις, από τις οδηγίες όπως ε, για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση των ιατρών. Ορισμένοι επίσης από τους ε, επαγγελματίες υγείας ε, ίσως είναι αυτοαπασχολούμενοι σε, ε, σε, σε, στον τομέα της υγείας και επομένως δεν εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές. Θα πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη στις αναγνωρίσεις. Βεβαίως οι σχετικές απαιτήσει δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο, φραγμό για την αναγνώριση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ξεκάθαρη μελέτη επιπτώσεων και η περιπτώσεις να κρίνονται αναπερίπτωση, όταν δηλαδή υπάρχει πραγματική προστιθέμενη αξία. Η κάρτα θα πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα για τους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή όμως ο επαγγελματίας διαθέτει την κάρτα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για την αρμόδια αρχή η αναγνώρισή της, να είναι υποχρεωτική η αναγνώρισή της. Μπορούμε να βασιστούμε στην πλατφόρμα IMI που είναι ε, ασφαλής αντί να αρχίσουμε με κάτι αντελώς καινούριο από την αρχή δηλαδή. Ευχαριστώ. Τούρινεν μεταξύ των συντονιστών. Θα μιλήσω όμως δανέζικα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση αποτελεί σωστή αφετηρία για την περαιτέρω εργασία μας και την ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα περισσότερα από τα όσα διαλαμβάνει η εκθεσή της. Όταν μιλούμε για ευκαμψία, για μείωση της γραφειοκρατίας, για σεβασμό της ε, ασφάλειας και της υγείας στο χώρο απασχόλησης, όταν μιλούμε για το ότι οι γλώσσες δεν πρέπει να αποτελούν φραγμό, Αυτά είναι σωστά και ιδίω για τους νεότερους υποψηφίους που έχουν και δικαίωμα σε ίση μεταχείριση. Αυτά, σε αυτά συμφωνώ. Υπάρχουν τώρα και τρία σχόλια που επιθυμώ να κάνω και που βρίσκω ότι είναι σημαντικά. Πρώτο, η συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη. Στην έκθεση εκφράζεται η ευχή, η επιθυμία, σχετικά δηλαδή με την ανάγκη προώθηση της ε, ε διαρκούς εξέλιξης, εγώ νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε και περισσότερο. Να τονίσουμε δηλαδή το δικαίωμα σε αυτήν, στην οδηγία, για πτυχές ασφάλειας στον τομέα της υγείας, καθώς και για την αύξηση του επίπεδου των προσόντων, που είναι σημαντικό. Το άλλο σχετικά με την μερική πρόσβαση. Δεν βλέπω κανέναν που να συμφωνεί ότι είναι καλή ιδέα. Εάν υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα, αν εμφανιστεί και α το πει, γιατί εγώ δεν το είδα ακόμη. Διότι αλλιώ για ποιο λόγο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την έννοια. α την εγκαταλείψουμε. Εκτός αν κάποιος επιμείνει ότι πρέπει να διατηρηθεί. Το τρίτο είναι τα σχετικά με τα προσόντα που βρίσκω ότι στενεύουν πολύ ορισμένα αντικείμενα στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχουν και ορισμένες παραδόσεις, ισχυρές παραδόσεις μέσα σε ε, χώρες μέλη, αλλά και εντός ορισμένων επαγγελματικών κλάδων, που είναι σημαντικό να γίνουν σεβαστοί. είναι σημαντικό να αντιληφθεί το Κοινοβούλιο ότι αυτά εδώ προωθούνται με συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων. Δεν θα πρέπει οι γραφειοκράτες των Βρυξελών να τα ρυθμίσουν τα πράγματα αυτά. Είναι σημαντικό αν θέλουμε να συνεχίσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Αυτά είναι σημαντικά, νομίζω, τρία αυτά θέματα. Κατά τα άλλα δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο και όπως είπα αποτελεί καλή βάση για την περαιτέρω εργασία μας. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ, καθώς επίσης ευχαριστώ όλους τους ε, σκιώδεις και σκιώδεις άλλοι που επιθυμούν να ομιλήσουν, η κυρία Γκέπχαρτ επίσης θέλει να προσθεθεί. Θα πω τα ονόματα τώρα. Παρακολουθώ λίγο και την ώρα, γιατί έχουμε και άλλα δύο θέματα. Mr. Juvin, Mr. Correa de Campos, Mrs. Corazza Bildt, Mrs. Weiler, Mr. Schwab, Mrs. Gephardt, and did, I, did, did Mrs. Irigoyen, I wasn't sure. No, okay. Is that anybody else? Κάποιος άλλος που θέλει το... Ναι, δεν, σας αποκλείω, αλλά θα ήθελα να μιλήσετε και εσείς επί του θέματος. Θα ήθελα να λάβετε το λόγο για δύο-τρία λεπτά το πολύ, όχι παραπάνω. Και ο κύριος ε, Τζόρνταν θα, θα κρατάει το χρόνο, έτσι ώστε να αρκεστείτε στο χώρο σας. Γουτιέρας Κορτίνεθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι συμφωνώ μαζί της και ιδίως ως προς τη στάση της, δηλαδή αναγνωρίζω τη στάση της και ταυτίζομαι με αυτήν. Θα ήθελα όμως να την υποστηρίξω έτσι ώστε να είμαστε πιο απαιτητικοί από το σύστημα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε ορισμένες ιδέες και όχι να μην είμαστε απαιτητικοί και πιστεύω αρχικά ότι ως προς την αναγνώριση των τίτλων και των προσόντων δεν πρέπει να τα διαχωρίσουμε διότι συμβαδίζουν. Διότι όλα εξαρτώνται από τους τίτλους και τα επαγγελματικά δηλαδή προσόντα. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο, γιατί νομίζω ότι ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, μία νοσηλεύτρια, καταρχήν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους τίτλους τους. Και ε, εάν δεν αναγνωριστεί ο τίτλος δεν μπορεί να δουλέψουν στη δημόσια διοίκηση. Αυτό τουλάχιστον ισχύει στην Ισπανία. Θα ήθελα λοιπόν η ενιαία αγορά να ε, ομιλούν για ένα δικαίωμα στην εργασία. Άρα ε, να πρέπει να υπάρχει ρύθμιση ή μη ρύθμιση αυτό να ισχύει. Και εάν δεν μιλάμε για τίτλους από κοινού με επαγγελματικά προσόντα τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Το διοικητικό σύστημα του κράτους τι κάνει πολλές φορές αρνείται τον τίτλο. Πολλές φορές δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κρατικό πρόσκαμα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ορίσουμε μία νέα ρύθμιση για τη ρύθμιση. Όσο λιγότερα προσκόμματα τόσο το καλύτερο. Δηλαδή ο τίτλος θα πρέπει καταρχήν να αναγνωριστεί. Μία νοσηλεύτρια είναι νοσηλεύτρια, ένας υδραυλικός είναι υδραυλικός και ούτω καθεξής. Αυτό προαπαιτεί η κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής ε, κατάρτιση, αλλά έχουμε να αναγνωρίσουμε μια εργασία, μια αγορά εργασίας. Πολλές φορές και από πίσω υπάρχουν τα συνδικάτα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές ε, φορές όταν μιλάμε ας πούμε για τέχνη θα πρέπει η ξεναγή, η ιστορική τέχνης να ε, δίνουν εξηγήσεις. Δεν θα πρέπει όμως να δεχτούμε, να δεχόμαστε ε, μεσαιωνικές συντεχνίες. Θα πρέπει να απαρνηθούμε αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι το σύστημα αναγνώρισης είναι ταχύτερο από την κρατική αναγνώριση. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ρύθμιση. Γιατί ο καταναλωτής ή ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει ποιος δεν δέχτηκε τον τίτλο του και γιατί δεν δέχτηκε τον τίτλο του. Ευχαριστώ πολύ. Σας έδωσα περισσότερο χρόνο γιατί είσαστε σκιώδης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και ε, αναμένουμε και την ε, απάντηση της κυρίας Μακλάρκιν σε σχέση με τα δεδομένα της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Ο κύριος Ζουβέν. Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η δυσκολία προέρχεται από το γεγονός ότι μία νοσηλεύτρια δεν είναι νοσηλεύτρια πολλές φορές. Δηλαδή όταν μία νοσηλεύτρια καταρτίζεται στο, έχει μία κατάρτιση στον Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχει την ίδια κατάρτιση όπως στην Αυστρία. Και πολλές φορές θεωρούμε ότι υπάρχει διαφορά. Εάν όμως υποστηρίζουμε αυτή τη διαφορά και στεκόμαστε αυτή τη διαφορά, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Σε 5, 10, 20 χρόνια θα έχουμε την ίδια συζήτηση. Γιατί έχουμε να κάνουμε με την αρχή της επικουρικότητας, όπου τα προγράμματα δεν καταρτίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικές καταρτήσεις. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι στον τομέα υγείας βλέπουμε ότι οι, οι ασθενείς διατρέχουν κίνδυνο, θεωρούν, όταν δεν έχουν την υποστήριξη του ιατρικού προσωπικού που δεν είναι από τη χώρα τους. Δηλαδή, ε, πολλές φορές ε, γνωρίζουμε ότι σε Αυστρία ή Γαλλία ή στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, οι νοσηλεύτρες έχουν άλλη ε, κατάρτιση. Μην λοιπόν δεχτείτε αυτό το θέμα ασφάλειας. Γιατί θεωρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία η υποστήριξη του συστήματος είναι ίδια, δηλαδή οι ασθενείς δεν διατρέχουν κίνδυνο. Το θέμα της επικουρικότητας λοιπόν θα πρέπει να το δεχτούμε υπάρχει και ένα 28ο πρόγραμμα, το οποίο δεσπόζει των εθνικό, Διότι οι εθνικοί εγωισμοί, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι μικροσυντεχνίες, τι μας λένε, κάθε φορά προβάλλουν το δικό τους πρόγραμμα στα κράτη τους, εξαιτίας αυτής της επικουρικότητας που μας έχει επιβληθεί. Ας προσπεράσουμε τη δυσκολία, διότι σε 10 χρόνια θα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να ε, επιβάλλουμε ένα 28ο πρόγραμμα, όχι ένα ελάχιστο πρόγραμμα, ένα 28 ο ε, πρόγραμμα δεν θα πρέπει να είναι ένα άλοθη, αλλά ένα πρόγραμμα που δεσπόζει τον 27 σε όλα τα επαγγέλματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, ε, διότι γνωρίζουμε ότι έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό τον ε, τομέα και ο κύριος Δεκάμπος έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο Μακλάρκιν για την εργασία της η οποία είναι ιδιαίτερα εκτενής και ασχολείται με όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Δηλαδή ε, μιλά για τον τομέα των εγγύσεων προς ε, όλα τα επαγγέλματα. Συμφωνώ μαζί της και με την πρότασή της σε σχέση με την τάχιστη μεταφορά των οδηγίων. Αν και θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αυτή η οδηγία μεταφέρθηκε τόσο αργά. Συμφωνώ επίσης με το σύστημα προειδοποιήσεων ότι το σύστημα είναι ιδιαίτερα φορτικό σήμερα με τα συστήματα online, τις νέες τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Όμως, έχω την εντύπωση ότι η πρόταση είναι κάπως περιοριστική, πιο συσταλτική είναι η ερμηνεία της σε σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων. Υπάρχει λοιπόν συσταλτική ερμηνεία ε, για, τις, για επαγγελματίε από τρίτες χώρες, έτσι ώστε να μην γίνεται forum shopping, γίνεται λόγος για μια κοινή πλατφόρμα, την οποία δεν γνωρίζουμε πολύ καλά, διότι δεν μας επιβλήθηκε αλλά εάν πραγματικά υπάρχει θα πρέπει να εποπτεύεται από το Κοινοβούλιο. Έτσι αναφέρεται, αυτό δεν το κατανοώ. Και υπάρχει μεγάλη δέσμευση στον τομέα και εποπτεία στον τομέα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Εάν μιλάμε για ιδιαίτερα θα πρέπει να αρχίσουμε από τον τομέα υγείας, μετά να περάσουμε στους πολιτικούς ε, μηχανικούς, στους δικηγόρους και ούτω καθεξής και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη στην αγορά από πλευράς επαγγελματιών, διότι υπάρχει καθαρά συντεχνιακή προσέγγιση και γι' αυτό άργησε να μεταφερθεί η οδηγία. Τα κράτη-μέλη θα ήθελα να υπάρχει ενιαία αγορά, περισσότερη ενιαία αγορά όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, επόμενη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά σας ξαναβλέπω ε, και χαίρομαι που αρχίζουμε έτσι καλά τη χρονιά. Συμφωνώ σχεδόν σε όλα με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και συμφωνώ και με την απλοποίηση ε, και ότι όσο γίνεται καλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Συμφωνώ και με την κυρία Βερνιό ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένα μηνύματα να στέλνουμε ε, στους Ευρωπαίους πολίτες ότι κάνουμε σημαντική δουλειά που τους αφορά και το θέμα της επαγγελματικής κάρτας να είναι προαιρετική. Συμφωνώ με την Κωνσταντς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω να προχωρήσουμε παρά το οικονομικό κόστος και τις τεχνικές ε, πτυχές. Ε, τα ζητήματα υγείας βεβαίως είναι από τα πιο περίπλοκα, αλλά θα ήθελα να θυμίσω ότι πέρυσι επιτέλους νομοθετήσαμε για την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και ε, ε της υγείας Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία και τμήμα αυτή είναι αναγνώριση των επαγγελματικών προσώνων. Και θα πρέπει παντού στην Ευρώπη να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε ιατρικό επάγγελμα, οποιοδήποτε επαγγελματία υγεία μπορεί να εγκατασταθεί σε μια άλλη χώρα τη Ένωση και να εργάζεται. Οπότε δεν χρειάζεται ένα επιπλέον σύστημα, αλλά να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία και τις πτυχές που χρειάζεται ε, να εναρμονίσουμε. Ευχαριστώ πρώτα. Βάιλερ. <clears throat> Η κυρία Μπίλτ δίκιο έχει. Έχουμε ήδη οδηγία. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να επαναπαυθούμε, διότι δεν εφαρμόζεται ορθά η οδηγία αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν με ακούτε τώρα. Δεν εφαρμόζεται ορθά η οδηγία. Διότι άλλως δεν θα είχαμε σήμερα το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής. Ούτε θα συζητούσαμε ποιες διορθώσεις πρέπει να επέλθουν και ποιες απλουστεύσεις. Ιδού λοιπόν πόσο παράδοξη είναι η συμπεριφορά ορισμένων επαγγελματικών οργανώσεων ορισμένων χωρών, διότι όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη ειδικευμένων, ε, ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, βρίσκονται γρήγορα τρόποι να ξεπεραστούν οι φραγμοί για τις αναγνωρίσεις όχι τόσο για τους γιατρούς, όπου έλλειψη υπάρχει πια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Για νοσηλευτές και νοσηλεύτριες επίσης δεν υπάρχουν σχεδόν προβλήματα, διότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες τέτοιου ειδικευμένου προσωπικού. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να καταστήσουμε τα μέτρα αυτά γενικά δεσμευτικά σε όλη την Ευρώπη. Αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συγγετριά μας μπορούν να αποτελέσουν έναν τρόπο, αλλά τα επιγραμμικά συστήματα και οι διάφορες επαγγελματικές κάρτες δεν αρκούν εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ίσως πρέπει λοιπόν οι χώρες μέλη να συζητήσουν με τους εθνικούς βουλευτές ή να συζητήσουμε και εμείς με τους εθνικούς βουλευτές να το κάνουμε αυτό με μια βίντεο διάσκεψη έτσι ώστε οι ίδιες χώρες μέλη να προχωρήσουν στην κατάργηση των φραγμών της κινητικότητας των εργαζομένων στους τομείς αυτούς. Νομίζω η Δανή συνάδελφος είπε πριν και το βρίσκω σωστό ότι οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές παραδόσεις. Για παράδειγμα στη Γερμανία έχουμε ένα δι, διητό σύστημα με ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Έχουμε το σύστημα αυτό κοινό με το Λουξεμβούργο και την Αυστρία για τους ε, ε, τεχνίτες. Τα βάλαμε αυτά μια χαρά στην πρώτη οδηγία και ουδέν, πρόκυ... Ε, ουδέν πρόβλημα προέκυψε. Δεν επιτρέπεται αυτά τώρα να ξεθεμελιωθούν με την δεύτερη οδηγία. Το γνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε τα όσα θετικά αποτελέσματα υπήρξαν από την πρώτη οδηγία να μην χαλάσουν τώρα με αυτήν εδώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σφάπ και μετά κύριε Κέπχαρτ. Ευχαριστώ. Δεν μένουν πολλά να πει κανείς, διότι καταρχήν συμφωνούμε όλοι. Νομίζω ότι οι έπαινοι που ακούστηκαν για την έκθεση της κυρίας Λάρκιν είναι ορθή και αυτό ισχύει για πολλά θέματα που διαλαμβάνει. Τονίζω ιδιαίτερα ότι η πρόταση σχετικά με την επαγγελματική κάρτα πρέπει να εξεταστεί βαθύτερα. Ποιο, ποια είναι δηλαδή η προστιθέμενη αξία που προσφέρει η κάρτα αυτή. Πάντως οπωσδήποτε να υποστηριχθεί και αυτό ισχύει και για το γεγονός ότι η κυρία Μακλάρκιν θεωρεί ότι ένα τέταρτο όλων των 800 επαγγελμάτων που έχουν μέχρι τώρα καταχωριστεί διαρωτώ με και εγώ αν είναι ανάγκη για παράδειγμα να ε, ρυθμιστεί το επάγγελμα του μπάρμαν ή μήπως εκεί είναι καλύτερα να αφηθεί κάποια ελευθερία. Επανεξέτασα τις σχετικές εκθέσεις και έχω μια πληροφορία. Δύο τρίτα, σύμφωνα με τη στατιστική του Solvit, όλων των προβλημάτων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων προέρχονται από τέσσερις μόνο χώρες μέλη. Και ίσως είναι απαραίτητο να εξετάσουμε γιατί προκαλούνται τόσα πολλά προβλήματα. Ρωτάει η κυρία Γκέπχαρτ, ποιε χώρε. Λοιπόν, κύριε, πολύ κύριε Γκέπχαρτ, ευχαρίστω να σα δώσω το έγγραφο που έχω, αν θέλετε. Μπορείτε να τα διαβάσετε μετά. Δεν θα ήθελα να τα πω τώρα προφορικά ποιε είναι οι χώρε αυτέ. Η κυρία Γκέπχαρτ, παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου επιθυμώ να επενέσω την έκθεση για το θετικό της περιεχόμενο. Παρά τα αυτά νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Θα ήθελα να δοθεί πολύ περισσότερη έμφαση στο ότι τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, με τις μέχρι τώρα οδηγίες δηλαδή, σχετικά με την ελευθερία δικινήσεως τουλάχιστον στα χαρτιά, ότι αυτός πρέπει να παραμείνει ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε ιδιαίτερα για τα ιατρικά και άλλα σχετικά επαγγέλματα, έχουμε μια αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση. Και ε, να αμφισβητηθεί αυτή, αυτό θα προκαλέσει πολλά προβλήματα, αφού έχει επιτευχθεί ένας αυτοματισμός. Νομίζω αυτό λείπει στην έκθεση, ότι θα πρέπει δηλαδή να τονιστεί πολύ περισσότερο. Και επίσης περισσότερη έμφαση να δοθεί στην ευθύνη των χωρών μελών, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. αναφέρεται στο θέμα αυτό σε κάποιες παραγράφους η κυρία Λάρκιν, αλλά νομίζω πρέπει να τονιστεί πολύ περισσότερο. Ότι δηλαδή τα όσα ζητούμε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τα όσα έχουν επίση εγκρίνει οι κυβερνήσει και τα εθνικά κοινοβούλια, να εφαρμοστούν πραγματικά και να τεθούν σε ισχύ, έτσι ώστε οι πολίτε αμφωτέρων των φίλων να μπορούν να υποφεληθούν από τι ρυθμίσει αυτέ. Αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει, όπως είπα, να τονίσουμε πολύ περισσότερο μέσα στην εκθεσή σας. Έχω ωστόσο και μία ερώτηση σε ό,τι αφορά τη μερική πρόσβαση. Όντως, καμιά φορά είναι απαραίτητο να υπάρχει μερική πρόσβαση και δεν το αμφισβητώ. Αλλά είναι δευτερεύον. Μερική πρόσβαση που θα ενισχυθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει σε κατακαιρματισμό πάλι και σε δυσχέρανση. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε αυτό το πράγμα που επιθυμούμε να βοηθήσει ορισμένα αποτελέσματα να μην οδηγήσει τελικά σε αντίθετα αποτελέσματα. Πλήρης πρόσβαση λοιπόν, όσο είναι δυνατόν αυτό, βεβαίως με τήρηση των προδιαγραφών με τήρηση των διατάξεων και υποφελία του ασθενού ή του καταναλωτού. Στην παράγραφο 8 αναφέρεστε και στα ρυθμισμένα αποτελέσματα. Όντω σε ορισμένε χώρε αυτά αποτελούν πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, η ρύθμιση είναι απαραίτητη, η κανονιστική ρύθμιση δηλαδή, για την εξασφάλιση τη ποιότητα. Και εδώ νομίζω πρέπει να εξετάσουμε λίγο προσεκτικότερα και να διατυπώσουμε προσεκτικότερα αυτό που λέτε με τη φράση σας ότι ο συνολικός αριθμός των ρυθμισμένων ε, επαγγελμάτων συγγνώμη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειωθεί. Ναι, αλλά πώς, με ποιο τρόπο, με ποια κριτήρια. Δεν μπορεί κανείς να το λέει αυτό ή να το γράψει στην έκθεση με τόσο γενικό τρόπο, διότι πολλά ρυθμισμένα επαγγέλματα είναι και η βάση για την οποία αμείβονται καλύτερα οι επαγγελματίε αυτοί. Ενώ το αντίθετο, η απελευθέρωση θα σημάνει και μείωση των αμοιβών των επαγγελματιών αυτών. Τέλος, η επαγγελματική κάρτα, που για μένα είναι σημαντικό. Ασφαλώς και κάτι τέτοιο, μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να είναι ελευθέρα επιλογή του επαγγελματία. Ουδής μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει την κάρτα αυτή. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσουμε με θετικότερο τρόπο την πρόταση αυτή. Και βεβαίως υπάρχουν ε, επιφυλάξεις και βεβαίως υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν, αλλά ας μην βάζουμε αυτές τόσο πολύ στο προσκήνιο, όσο την συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία που θα προκύψει. Όπου υπάρχουν δηλαδή ήδη ε, ευρωπαϊκά αναγνωρισμένες επαγγελματικές κάρτες που σημαίνουν ελευθερία προσβάσεως, αναγνωρισμένη από τις ε, εθνικές αρχές, αυτό είναι που θέλουμε να επιτύχουμε εν τέλει τα θέματα λεπτομεριών, δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί η ρύθμιση αυτή, με ποια κριτήρια και ούτω καθεξής, αυτά θα πρέπει να είναι δευτερεύοντα εν προκειμένου. Εδώ, στην έκθεση πρωτοβουλίας που συζητούμε, δεν είναι στην νομοθετικού περιεχομένου, είναι περισσότερο μια κατάθεση της πολιτικής μας βούλησης. Άρα, ας μην προτάξουμε κυρίως τα προβλήματα, ας εξηγήσουμε ποιους στόχους θέλουμε να επιτύχουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους και όλους για την συμβολή σας στη συζήτηση που πρόσφερε πολλές θετικές ιδέες. Θα παρακαλέσω τώρα την Επιτροπή να λάβει το λόγο, να εξηγήσει τι έχει γίνει με τις διαβουλεύσει κλπ. Και τον ευχαριστώ και για την ε, θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ε, στις, ε, στους εκπροσώπους μας στις ομάδες εργασίας. Που αυτά προκύπτουν ως ωφέλη από τη νέα ε, συμφωνία πλαίσιο. Αυτά ήθελα να τα τονίσω και δημοσία, όπως αντιληφθήκατε. Λοιπόν, κύριε Τίτσερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την συγκεκριμένη Είναι πάρα πολύ σαφής ε, και συγκεκριμένη έκθεση για ένα θέμα περίπλοκο. Δεν θα εξαντλήσω ένα πεντάλεπτο που μου δίνετε. Θα είμαι ε, σύντομο. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πράσινη βίβλο. Δεν έχουμε λάβει λοιπόν οριστική θέση και βεβαίω θα ακούσουμε προσεκτικά αυτό που θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση πρωτοβουλία ε, προς την Πράσινη Βίβλο. Θα ήθελα να θυμίσω, μου επιτρέπετε, ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι τμήμα τη ε, ε, πράξης αγοράς. Και δύο είναι τα κίνητρά μα εκεί. Πώς μπορούμε να τονώσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Άκουσα ε, πολλά για τη δημόσια υγεία, για την ασφάλεια που είναι σημαντικά για τους πολίτες. Ωστόσο υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο εξίσου σημαντικό για μας και λίγο πιο δύσκολο που είναι η ανάπτυξη οικονομίας μας. Εκεί επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθεί η οικονομία, πώς θα βγούμε από την κρίση του ευρώ που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Και με βάση αυτά τα δεδομένα θα ήθελα να κάνω δύο μόνο σχόλια. Το ένα αφορά την παράγραφο 4 για τις ε, προσωρινές υπηρεσίες και την περιστασιακή παροχή τους. Βεβαίως, ε, πριν από τέσσερα χρόνια σε Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε ότι θα απεμπολίσουμε την πρώτο, τον πρώτερο έλεγχο των προσόντων με μόνη εξαίρεση τα επαγγέλματα δημόσιας υγείας και ασφαλείας. Αυτό το λέει και η οδηγία. Τι άλλο ε, θα πρέπει τώρα να διευκρινίσουμε. Ανισχούμε λίγο, μην ξανανοίξει η συζήτηση που έχει γίνει ήδη για την προηγούμενη οδηγία. Το 2002 έκανε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισχύουσα οδηγία, εισάγοντας αυτή την έννοια. Ε, ε, με ένα ε, νομικό, μια νομική παραδοχή ότι χρειάζονται λίγες μέρες και τελικά ε, οδηγηθήκαμε σε μεγάλη αποτυχία και ε, αποφάθηκε το δικαστήριο. αλλά το δικαστήριο λέει θα πρέπει κατά περίπτωση να αποφασίζουμε και αυτή είναι η νομολογία. Τώρα χρειάζεται να ανοίξουμε συζήτηση για μια προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών. Είναι καλό για την οικονομία μας. Θέλουμε και άλλους κανόνες. Χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες εκεί. Αναφερθήκατε ιδιαίτερα ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία των καταναλωτών που πηγαίνουν σε άλλη χώρα. Το σημειώνω αυτό, αλλά κατά τα άλλα ισχύει κάτι για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω και πάλι με ε, γνώμονα την ε, ανάπτυξη οικονομίας είναι αυτό το θέμα της περιορισμένης πρόσβασης. Ναι, το καταλαβαίνω ότι η μερική πρόσβαση είναι κάτι που ενοχλεί τους επαγγελματίε. αλλά αυτό δεν είναι έμπνευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μήπω χρειάζεται λοιπόν διευκρίνηση εδώ. Η αφιτηρία ποια είναι. Έρχεται κάποιο από τη χώρα του, πηγαίνει σε άλλη χώρα, ε, ασκεί μια οικονομική δραστηριότητα και θέλει να την ασκήσει σε μια άλλη χώρα. Και ε, σε ό,τι αφορά το σημείο 13 λοιπόν, δεν αφαίρεστε μόνο σε επαγγέλματα υγείας, αλλά και άλλα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσει στην ασφάλεια. Κοιτάξτε τι έχει πει το δικαστηρίο ε, για ε, τους μηχανικούς και για άλλους τομείς. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το θέμα, αλλά πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Ανά περίπτωση λοιπόν αντιμετωπίζουμε όταν υπάρχουν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, στη συνέχεια τα κράτη-μέλη αν χρειαστεί προσαρμόζουν τους κανόνες για το συγκεκριμένο επάγγελμα, όχι εγκάρσεις ε, ρυθμίσεις. Τέλος για την επαγγελματική κάρτα. Ε, έχει δίκιο στις προτάσεις εισηγήτρια, ισχύουν όλες. Ξέρετε ότι θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό στο Φόρουμ για την Εσωτερική Αγορά αρχές Οκτωβρίου. Εργαζόμαστε ε, στα τεχνικά ζητήματα εμπειρογνώμονες και σας ε, προτείνω, σας προσφέρω αν θεωρείτε χρήσιμο μέχρι τότε να έχετε και άλλες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε στη διάθεσή σας, πρόθυμοι. Σας είπα ότι είναι ομάδα εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι το σωστό φόρουμ εκεί. Εγώ αυτό σας προσφέρω να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση πριν ε, τη διεξαγωγή. Τελικά μίλησα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Μακλάρκιν, ε, για να συνοψίσει και να κλείσει και να επαναλάβουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ, εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Γνωρίζω ότι ε, έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ όλους και όλες τις ε, σχιώδεις που με βοήθησαν ιδιαίτερα με τα δεδομένα που μου έδωσαν και ελπίζω να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες όλων των πολιτών και καταναλωτών ως προς τις προτεραιότητες για την ενιαία αγορά στην Επιτροπή αυτή και διαμέσου αυτής της έκθεσης πρέπει να πούμε στην Επιτροπή τι σκεφτόμαστε και να αντικατοπτρίζουμε τις απόψεις των ε, διαβουλεύσεων για να δείχνουμε ότι εισακούονται οι προσδοκίες των επαγγελματιών και των πολιτών. Όταν μιλάμε για προσωρινή πρόσβαση, ξέρω ότι υπάρχει απόφαση του 10, αλλά όπως είπατε, οι διαβουλεύσεις, η ανταπόκριση στις διαβουλεύσεις δείχνει ότι δεν χρειάζεται ε, αυτή η οδός, να ακολουθήσουμε αυτή την οδό από πλευράς νομικής προσέγγισης, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πού θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση σε αυτήν την οδηγία, αλλά το θέμα κλειδί είναι η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει να επιβλέπουμε επίσης την κατάσταση, να υποπτεύουμε την ε, κατάσταση ως προς την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, τη μεταφορά στην εθνική ένωμη τάξη, έτσι ώστε οι κατανοτές να έχουν την προστασία που επιβάλλεται και οι επαγγελματίε να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα σε πρεχόμενο στάδιο, όταν δηλαδή φτάσει το θέμα στο Συμβούλιο. Προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα. Σε σχέση με τους σκιώδεις, θα ήθελα να γνωρίζουν οι σκιώδεις ότι θα έχουμε δύο ε, συνεδριάσεις το Σεπτέμβριο τώρα ε, στο Στρασβούργο και στις δύο συνόδους και κύριε Τίτσερ αν θέλετε μπορείτε να παρευρεθείτε σε μία από τις δύο συναντήσεις. Θα δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμούς. Αναμένω τις ε, τροπολογίες σας μέχρι την προθεσμία της 17ης δηλαδή. Επίσης θα ήθελα να επιβεβαιώσω το ότι στις 19 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μία νέα τηλεδιάσκεψη με την ομάδα εργασίας της ε, Bundestag στις 5.30. Δεν ξέρω ποιοι ε, σε ποια αίθουσα. Γι' αυτό θα θέλαμε όλοι οι σκιώδεις να παρευρίσκονται σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, διότι και από πλευράς Bundestag θα υπάρχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα παρευρίσκονται όλοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι της ομάδας εργασίας. Στο 2Q2 θα γίνει η τηλεδιάσκεψη που είναι μεγαλύτερη αίθουσα στο δεύτερο όροφο στις 5.30 της 19 Σεπτεμβρίου και μετά θα ψηφίσουμε στις 17 Οκτωβρίου στην Επιτροπή την έκθεση Μακλάρκιν και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Θα έχουμε δηλαδή επαρκή χρόνο έτσι ώστε να έχουμε και την πρόταση της προτάσης της Κομισιόν που περιμένουμε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ή λίγο μετά γύρω από εκείνη την χρονική περίοδο, κύριε Τίτσα, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ όλους. Περνάμε στο επόμενο θέμα. ως προς το προσχέδιο έκθεσης που καταρτίστηκε πριν από το καλοκαίρι και θα εξετάσουμε τώρα όσοι ε, θέλουν μπορούν να αποχωρήσουν. Το πρώτο σχέδιο, γνωμοδό, το σχέδιο γνωμοδότησης αυτό αφορά ένα σχέδιο προς την ε, ΙΜΚΟ, η οποία έχει και μία, συντάσσει μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, um, την Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου, με συγχωρείτε. Έχουμε την κυρία Πέντε Γκάσλα Χαγκάρτ, Κάμφε, η κυρία Ρούλερ δεν μ' ακούει. Εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μιλήσει και από τους ε, πρασίνους και εγώ είμαι σκιώδης και γι' αυτό θα έχω τη δυνατότητα να λάβω το λόγο. Δίνω το λόγο στην κυρία Λεγκρίπ τώρα για το σχέδιο γνωμοδότης αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα των φραγμών στις συναλλαγές της επενδύσεις. Το Μάρτιο η Επιτροπή είχε συντάξει μία έκθεση για τα εμπόδια στις συναλλαγές και τις επενδύσεις για να δούμε ποιες δράσεις θα μπορούσαν να προβληθούν έτσι ώστε να αρθούν τα εμπορικά προσκόμματα που δεν είναι δασμολογικής φύσης και που αποτελούν πραγματικό φραγμό ως προς εμπορικές συναλλαγές. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της Κομισιόν, η οποία είχε προανακοινωθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Δεν μιλάμε λοιπόν για τη μείωση των δασμολογικών φραγμών πλέον, αλλά και για την άρση των ρυθμιστικών φραγμών. Το ίδιο ακριβώς τονίζει και η Κομισιόν διότι έχει μεγάλη σημασία για τους, ως προς τους στρατηγικούς μας επενδυτές Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Αργεντική, Αργεντινή, Ρωσία και ΙΠΑ. Ε, εκτός Αργεντινής και Βραζιλίας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ε, διμερείς, ε, ε, διμερείς συμφωνίες συναλλαγών. Όπως ξέρετε, θα υπάρχει μάλλον μία έκθεση επιτροπής την οποία σας καλώ να διαβάσετε. Μιλάμε λοιπόν για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πρόσβαση προς τις αγορές των στρατηγικών μας εταίρων, έτσι ώστε να υπάρχει αμοιβαιότητα, να εποπτεύουμε το καθεστώς και να επαγρυπνούμε έτσι ώστε να μην υπάρχει προστατευτισμός δηλαδή να ε, μην προδικάσουμε αρνητικά αυτές τις ε, εμπορικές συναλλαγές. Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,5% εάν υπάρξουν ε, συγκεκριμένες εξελίξεις στους μη δασμολογικούς φραγμούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή μία οικονομική ανάπτυξη Αυτό αφορά και την πρόσβαση στις ε, δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει να υπάρχει διαρκής ε, προμήθεια στον τομέα αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θέμα των γεών και το θέμα των σπανίων ορυκτών από πλευρά των συναλλαγών μας με τις Κίνες και να λάβουμε υπόψη και τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις. Η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες από πλευράς όλων των αντιπροσωπιών καθώς και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών για να έχουμε μία ενιαία φωνή έναντι των εμπορικών μας εταίρων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να άρουμε αυτούς τους ε, φραγμούς του εμπορίου και των συναλλαγών. Η ίντα θα αποφανθεί επί της ουσίας και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στις δικές μας αρμοδιότητες. Υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών έτσι ώστε να άρουμε τα προσκόμματα που δεν έχουν δασμολογικό χαρακτήρα και να υπάρχει προσβασιμότητα στις αγορές. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ρυθμιστική προσέγγιση και στα πλαίσια της ΙΜΚΟ μιλήσαμε για αυτά τα ειδικά φόρα όπου συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η στρατηγική μας ΕΤΕΡ. Δηλαδή το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, εκεί όπου ορίζονται οι εταιρικέ σχέσεις και θα πρέπει να διευρυνθούν τα δεδομένα και να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Ως προς τις δημόσιες προμήθειες το συζητούμε στα πλαίσια της έκθεσης Ρούλε για την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων προμηθείων πρέπει να διανύσουμε ε, ένα πολύ μεγάλο ε, δρόμο μέχρι να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Όπως και από τον Επίτροπο Μπαρνιέ, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα και αμοιβαιότητα μέσα στα πλαίσια του ανοίγματο των αγορών δημοσίων προμηθειών. Και αναμένουμε και την προσαρμογή αυτού του μέσου και από την Επιτροπή, ιδιαίτερα στη, ως προς τις σχέσεις μας με την Κίνα. Θα πρέπει και εμείς να προσδώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα, διότι η Κίνα θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για την πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες. Επίσης προσδίδουμε μεγάλη σημασία στον διάλογο και τη συνεργασία με τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους και εδώ προσδίδουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προϊόντων και το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δύο θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει επί μακρόν. Η γνωμοδότηση είναι αυτή που βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι είναι μια βραχία έκθεση, περιμένω τη δική σας συνεισφορά και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σαφή επεξήγηση. Είναι πολύ καλή αυτή η έκθεση. Παρακολουθούμε και το βασικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Ας γίνει ένας γύρος λοιπόν. Η κυρία Πέντεγκάρντ έχει το λόγο. Καταρχήν είναι η πρώτη της έκθεση ως κοιόδης από πλευράς σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την Κωνστάς Λεγκρίπη για το σχέδιο γνωμοδότησής της. Βεβαίως είναι σημαντικό το στοιχείο της αμοιβαιότητας και των ε, ίσων όρων παιχνιδιού και την πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες, αλλά με σαφείς κανόνες. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας στάση και θέση απέναντι σε βασικούς εμπορικούς εταίρους. Αλλά γιατί να ξεχωρίσουμε την Κίνα ως, ε, μεταξύ των χωρών ας πούμε, που βάζουν εμπόδια ε, στις διαδικασίες δημοσίων έργων. Θα πρέπει γενικότερα να αναφερθούμε στους εμπορικούς εταίρους μας. Γιατί είναι μεγάλες οι εμπορικές ροές και ε, σε άλλους στρατηγικούς τομείς. Το 2011 είδαμε την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους φραγμούς και τα προβλήματα. Και οι αναπτυγμένες χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή έχουν διαπραγματευτεί περιορισμούς και καλύπτουν τις περισσότερες ε, περιπτώσεις και αγορές δημοσίων έργων. Από πλευρά μας και επειδή συμμετέχω στην αντιπροσωπεία για τις Ηνωμένε Πολιτείε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα των προδιαγραφών και των κανόνων. Συνδυασμένες αγορές, αλλά θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια. Πρόκειται για 122 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, χρησιμοποιεί εμάς που είμαστε στις αντιπροσωπείες και κοινοβουλευτικές επιτροπές με άλλες χώρες, να μας δείχνει ε, τα στοιχεία, να μας δίνει την πραγματογνωμοσύνη της για να μπορούμε να ε, εργαζόμαστε στον τομέα αυτό. Και επίσης ό,τι αφορά το εμπόριο και την αηφόρο ανάπτυξη, προστασία των κοινωνικών και των εργασιακών προδιαγραφών και στην Ένωση και αλλού σε παγκόσμιες αγορές, βλέπουμε ε, να ε, ε, διαβρώνονται, να μειώνονται οι προδιαγραφές και τα πρότυπα και αυτό να έρχεται και εις βάρος μας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που επανέρχομαι και εγώ μετά τις έννοιες διακοπές και βλέπω ότι ακολουθούμε τη γραμμή εκεί που την είχαμε αφήσει πριν το καλοκαίρι. Σε περισσότερα θέματα για το διεθνές εμπόριο Επ' αυτού ευχαριστώ την εισηγήτρια της συντάκτης νομοδότησης. Συμφωνώ ε, με τα όσα λέει σε πολλά σημεία που εγγράφονται και στη ε, γραμμή της δικής μου γνωμοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνας που θα συζητήσουμε αύριο. Αν μου επιτρέπετε ωστόσο μερικά σχόλια. Έχω μια ερώτηση για ένα από τα θέματα της νομοδότησης, που είναι και θέμα ε, του τίτλου. Οι επενδύσεις, γιατί εγώ αναφέρω πολλούς τομείς στη γνωμοδότησή μου, αλλά νομίζω ότι οι επενδύσει χρειάζονται ξεχωριστή και βαθύτερη προσέγγιση. Έχω μιλήσει με πολλούς εμπειρογνώμονε κατά τη διάρκεια τη σύνταξη τη δική μου γνωμοδότηση. Και το θέμα των επενδύσεων θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά ως παράγραφος στη γνωμοδότηση αφού ε, γράφει και ο τίτλος. Στο άρθρο 2, αν δεν απατώμε, γίνεται ειδική αναφορά και παραθέτω. Εύχεται η διαρθρωμένη διάλογοι επί τον κανονισμό που έχουν δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με ορισμένου από του εταίρου μα. Γιατί ορισμένου, έχετε υπόψη σα ε, συγκεκριμένη χώρα ή χώρε. Και αν ναι, πειράζει να τις κατονομάσουμε είναι γλωσσικό λάθος, έχει παρισπρίσει εδώ, ε, πρόκειται για συγκεκριμένες χώρες. Δεν ξέρω αν είναι ε, λεπτομέρεια, θα παρακαλούσα να μου τη διευκρινίσετε. Γενικά συμφωνούμε όλοι με τα θέματα που αναγράφετε στη γνωμοδότησή σας και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε θέλει να μιλήσει από την πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την πρότασή της. Υποστηρίζω κυρίως το δεύτερο σημείο που μιλάει για τις διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα και ε, είναι πολύ σημαντικό για μας. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο σημείο 4, το γράφει και δική μου έκθεση και χρειάζεται σε μεγαλύτερο βάθος συζήτηση ε, στην Επιτροπή. Γιατί στις δημόσιες αγορές βεβαίως και στις αναθέσεις θα πρέπει να σκεφτούμε τα εξή. Υπάρχει μια οδηγία βέβαια που ε, επιτρέπει όταν είναι ιδιαίτερα χαμηλές οι προσφορές ε, να απορρίπτονται. Τα κράτη-μέλη δεν το εφαρμόζουν και είναι ζήτημα αυτό και θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν το κάνουν. Αλλά δεν ξέρω εάν χρειάζεται επιπλέον ε, κανόνας ή άλλη νομοθεσία αφού δεν χρησιμοποιείται και δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα. Και στο θέμα της ανάθεσης των δημοσίων έργων, πολύ συχνά ποντάρουμε σε ε, ζητήματα που κινδυνεύουν να είναι προστατευτικά. Μήπως είναι εις βάρος μας αυτό. Κατανοώ ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε ε, σοβαρά ποια είναι τα μέσα εκείνα που ενδείκνυται και είναι και τα σωστά. Και ένα τελευταίο, το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει επιβάλει με ιδιαίτερα περιοριστικό τρόπο τη συμφωνία, δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα κάνουν και οι άλλες χώρες. Η επεξεργασία της οδηγίας νομίζω θα ε, μπορούσε να οδηγήσει σε ένα άλλο συμπέρασμα, να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στον εαυτό μας, να είμαστε λιγότερο αυστηροί και περιοριστικοί εδώ, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης το εξής. 1,3% των δημοσίων έργων είναι ε, πραγματικά έργα που έχουν διασυνοριακή σημασία. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα γραφειοκρατικά και οι περιορισμοί έχουν ιδιαίτερο νόημα. Ευχαριστώ. Να πω κι εγώ μερικά λόγια. Γιατί είμαι κι εγώ σκιώδης η γνωμοδότηση της κυρίας Λεγκρίπ. Γενικά συμφωνώ με το γεγονός ότι είναι πολύ καλό το πλαίσιο, αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι και ε, θα ενισχύσουν πολύ τη γνωμοδότηση. Ιδιαίτερα έχει δίκιο η κυρία Πέντεργαστ που λέει ότι δεν θέλουμε να κατονομάζουμε την Κίνα στα δημόσια έργα, στις δημόσιες αγορές και συμβάσεις. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω είναι πολύ αφελής. Και ε, ε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο κλειστή είναι η αγορά στις ΗΠΑ για τις δημόσιες προμήθειες. Εγώ ως μέλος Επιτροπής ε, και της Αντιπροσωπείας για την Ιαπωνία έχω μεταβεί στην Ιαπωνία και είναι πολύ κλειστή η αγορά τους για τις δημόσιες προμήθειες και θα μπορούσε να υποφεληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Και ε, ιδιαίτερα ε, μπορούμε να συνεισφέρουμε και με βάση τα όσα είπε η κυρία Ρούιλε από την εμπειρία της. Και θα πρέπει να δούμε και στις τεχνικές προδιαγραφές ε, το πρόβλημα, ότι δεν είναι ε, πάντα αντίστοιχοι οι ε, κανόνες που ισχύουν, ε, τεχνικές προδιαγραφές είναι επιπλέον εμπόδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα και στην Ιαπωνία όπου οι ευρωπαϊκές δοκιμές δεν γίνονται δεκτές και ζητούν και άλλες τεχνικές δοκιμές κτλ. Ε, όλα αυτά είναι φραγμοί μη τελωνιακοί ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν οπωσδήποτε και πολλές φορές... Ε, δεν υπάρχουν καθόλου επιστημονικά στοιχεία για ιδιαίτερους τομείς όπως είναι ε, η υγεία ή τα τρόφιμα ή τα ιατρικά μηχανήματα που κυκλοφορούν με ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν και αντίστοιχε προδιαγραφές και δεν τα δέχονται άλλες χώρες. Πάρα πολύ κρίσιμα αυτά τα θέματα και η κυρία Λεγκρίπ μιλάει για πρότυπα και για προδιαγραφές. και θα ε, συνεχίσει την προσπάθεια αυτή η κυρία αλλά πραγματικά τα πρότυπα και οι προδιαγραφές είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε και, να το συζητήσουμε στην Επιτροπή μας. Έχει δίκιο ο κυρία Λεγκρίπ. Βεβαίως εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, αλλά χρειάζεται να γίνει πρόοδος στη συνεργασία με τους Αμερικανούς, να έχουμε κοινά όργανα που να αντιμετωπίζουν ε, τις προδιαγραφές σε νέους τομείς, σε αναπτυσσόμενες περιοχές, ε, τομείς ή στην ανοτεχνολογία, στα ηλεκτρικά οχήματα, σε αναδυόμενους τομείς λοιπόν της οικονομίας, να μην εφευρίσκουμε τώρα νέα εμπόδια και νέους φραγμούς εμπορίου στις νέες τεχνολογίες. Πράγμα που συμβαίνει αυτό το γέρο. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες και να δείξουμε παγκοσμίω ότι έχει νόημα να επεξεργαζόμαστε παγκόσμια πρότυπα και να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή και η Κίνα και η Ιαπωνία. Νομίζω αυτό θα ήταν ένα καλό παράδειγμα για να προχωρήσουμε και εκ των προτέρων να λύνουμε τα προβλήματα, αντί να ερχόμαστε εκ των υστέρων που έχουν εδρεωθεί πολύ γραφειοκρατικά και είναι βαριές οι διαδικασίες. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε και τα τελωνία, γιατί εμείς είμαστε αρμόδιοι και η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εξαιρετική και εντοπίζει ακριβώς εμπόδια γραφειοκρατικά τελωνιακά για την εισαγωγή αγαθών, για τις ελέγχους στο τελωνία και αυτό είναι ένας νέος φραγμός. Τελειώνω λέγοντας ότι ε, καλό θα ήταν να πούμε κυρία Λεγκρίπ ε, ότι μπορεί να είναι θέματα διεθνούς εμπορίου αλλά την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνική γνώση την έχουμε εμείς που είμαστε Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Γιατί εργαζόμαστε σε εσωτερικό επίπεδο ε, για τέτοιους φραγμούς ε, επενδυτικούς, τεχνολογικούς, ε, διαφορετικές τεχνολογικές, τεχνικές προδιαγραφές κτλ. Και έχουμε εργαστεί πολύ σε αυτούς τους τομείς Ορισμένοι που είμαστε ακόμα μέλη εδώ και θυμάμαι ένα παλιό επίτροπο, το Πασκάλ Λαμι για θέματα εμπορίου που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία εσωτερικής αγοράς. Οπότε πιστεύω ότι και η δική μας Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής μας θα πρέπει να συμμετέχουν πολύ περισσότερο και πιο στενά να συνεργάζονται με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Και χαίρομαι που ε, παρευρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήρθε και ο Επίτροπος Επίσημα δεν συμμετέχουμε. Εγώ είμαι μέλος ε, ε, της Διευθυντικής Επιτροπής για το ε, διατλαντικό εμπόριο και αλλά θα κάνουμε να ζητήσουμε από την αντιπροσωπεία για τις Ηνωμένε Πολιτείε και τους συναδέλφους Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου να συνεργάζονται μαζί μας γιατί έχουμε γνώση, μπορούμε να βοηθήσουμε και θα βρούμε δρόμους να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν ξέρω, κάπως έτσι ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε σίγουρα ο συνάδελφος Βίτα Μωρέ που είναι ε, ο ομόλογο μου, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Διεθνού Εμπορίου, θα συμφωνήσει με αυτά. Αυτά ήθελα να πω εγώ ω και ο διηγητή. Άλλος συνάδελφος θέλει το λόγο. Ο κύριο Φαπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιορίσω σε τρία σχόλια. αφού συγχαρώ πρώτα την κυρία Λεγκρίπ για τη γνωμοδότησή της, που αποτελεί ένα καλά ισορροπημένο συνδυασμό των διαφόρων επιχειρημάτων, που είναι όλο και πιο σημαντικά για την Επιτροπή μας εν ώψη της παγκοσμιοποίησης, και τα όσα είπε ο Πρόεδρος σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν αποτελούν μια απλή απήχηση των όσων έχουν δεχθεί κατά επανάληψη, αλλά μας οδηγούν και να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Επιτροπή για να ενισχύσουμε και να κάνουμε πιο αποτελεσματικό τον διατραντικό αυτόν διάλογο. Μέχρι τώρα δεν έχουν επιτευχθεί πολλά στο πλαίσιο αυτό. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο η Επιτροπή μας να κάνει περισσότερα πράγματα. Δεύτερο, η Κίνα δεν θα έπρεπε να μπει στο επίκεντρο της εκθέσεως της κυρίας Λεγκρίπ. Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά για την ενιαία αγορά. Αναφέρθηκαν στην τυποποίηση, εγώ προσθέτω την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατάργηση φραγμών ε, στην πρόσβαση για τις αγορές και τα όσα είπε Ρούλε για την παράγραφο 4 δηλαδή, όπου είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη η διατύπωση και όντω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη κανονιστική ρύθμιση. Αλλά η υφιστάμενη συμφωνία, αυτό το General ε, Procurement, procurement εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις, αλλά δεν είναι σαφές ποιος μπορεί να προβάλλει τις επιφυλάξεις αυτές. Οι χώρες μέλη, η Ένωση και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να πούμε ωστόσο ότι αυτά αποτελούν μέρος ε, της, ε, του, του πλαισίου των δημοσίων αγορών των δημοσίων προμηθειών δηλαδή. Αυτά πρέπει να συζητηθούν εν προκειμένου. Και επειδή μιλήσατε και για την, το άνοιγμα της αγοράς στην Ιαπωνία, στις 8 Ιουλίου έγινε μια συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι η Ιαπωνία έχει ανοίξει μονάχα το 25% της ε, αγοράς της δημοσίων προμηθειών ο Καναδάς μονάχα το 4%. Βεβαίως δεν είναι και σαφές πώς προκύπτουν αυτά τα νούμερα. Θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει πώς προκύπτουν οι αριθμοί αυτοί. Πάντως, όπως είπα, θεωρώ ε, χρήσιμη την ε, έκθεση της κυρίας Δεγκρίπ. Σας ευχαριστώ, ε, ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους. ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει απόψεις. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που έχει προσφέρει με την έκθεσή της μια καλή βάση για την ανάπτυξη της ε, στρατηγικής μας. Η αφαίρεση αυτών των κολλημάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε την ετήσια έκθεση για τα κολύμπατα σε επενδύσεις και πρόσβαση στις αγορές. Θα συζητηθούν αυτά στο Εαρινό Συμβούλιο. Μπορούμε να κάνουμε και τη σύγκριση έτος προς έτος. Μια σύντομη παρατήρηση για την παρούσα έκθεση. Πρόκειται για θεμελιώδη ε, λίθο για τις σχέσεις μας δηλαδή με τρίτες χώρες, για την αξιοπιστία μας πώς επιβάλλουμε, πώς εφαρμόζουμε μάλλον τις ε, συμφωνίες εμπορίου, πώς παρακινούμε τις χώρες μέλη να συνεργαστούν στους δημιουργεί διαλόγους τους και με τρίτες χώρες και η αφαίρεση των κολλημάτων στο εμπόριο είναι υψηλής προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή σας και που το ενδιαφέρον αυτό το εκφράζει με έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την αφαίρεση των φραγμών στις ε, επενδύσεις και στο εμπόριο. Ενισχύεται τις, προ... τις... τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι σε μια προσπάθεια αφαίρεσης όλων των ειδών φραγμών, έτσι ώστε το διεθνές εμπόριο να γίνεται σε βάση ίσων όρων ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ο κ. Σφάπ έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ίσως μπορείτε να το σημειώσετε και να μας απαντήσετε έστω και γραπτός. Πάντως, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη ορισμένων από τα θέματα που ε, θέσατε και η κυρία Λεγκρίπ τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρωτίστως όλους τους παρεμβάντες, ιδίως τους σκιώδης για τις πολύ συγκεκριμένες και ακριβείς προτάσεις τους. Γνωρίζω ότι η βραχύτητα των προθεσμιών που αντιμετωπίζουμε δεν επέτρεψαν την τέλεση συνεδριάσεως με τους σκιώδεις πριν από την διακοπή των εργασιών μας και ναι μεν τα είπαμε με ηλεκτρονικά ταχυδρομεία αλλά και με την βοήθεια των συνεργατών μας. Ωστόσο δεν μπορέσαμε να προβούμε σε πραγματική ανταλλαγή απόψεων πρόσωπο με πρόσωπο. Και για το λόγο αυτό, στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως που σας υπέβαλα σήμερα, έχω αυτοπεριοριστεί σε ορισμένα θέματα, καθώς επίσης σε ένα μήκος κειμένου που είναι λιγότερο από το επιτρεπόμενο, έτσι ώστε να αφήσω χώρο για να εντάξω και προτάσεις και τροπολογίες ή άλλες παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία, ίσως όχι εξαντλητικά, πάντως ο διάλογος θα συνεχιστεί ιδίως με τους σκιώδεις σε μία συνεδρίαση που θα συγκαλέσω. Θα ήθελα να πω πρώτα να αναφέρω μια σημειολογική, αν θέλετε, παρατήρηση στην παράγραφο 2, όταν αναφέρομαι στον διαθρωμένο κανονιστικό διάλογο, στα, στον διαθρωμένο διάλογο σχετικά με τις προδιαγραφές, ορισμένοι από τους εταίρους μας, προτείνω μάλλον το διάλογο αυτό επειδή δεν υπάρχει τέτοιος διαθρωμένος διάλογος με ορισμένους το σύνολο μάλλον των εταίρων μας. και δεν έχω αναφέρει έτσι, δεν έχω απαριθμίσει όλους τους εταίρους. Είναι κάπως ασαφές και είμαι διατεθειμένη να κάνω τη σχετική διόρθωση και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χειριστούμε καλύτερα τις συνθήκες αυτού του διαλόγου είναι ίσως κάπως ε, σημειολογική παρατήρηση όπως είπα αυτό, ίσως και μετάφραση να μην απόλυτα ακριβή. Πολλοί από τους κοιόδης αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5 και το γεγονός ότι αναφέρομαι στις εμπορικές σχέσεις μας με την Κίνα. Εδώ θα προβώσω ορισμένε ορισμένες διευκρινήσεις. Όχι, δεν έχω καμία μανία με την Κίνα, βεβαίω είναι η δεύτερη δύναμη στον κόσμο και επομένως πολύ σημαντικός εταίρος. Δεν είναι ένας εταίρος από πολλούς. Είναι και μεγάλη ε, η βαρύτητα της Κίνας πλέον ε, στο διεθνές επίπεδο. Η Κίνα άλλωστε αυτή τη στιγμή προχωρεί σε μια προκτακτική φάση διαπραγματεύσεων για να ενταχθεί στην ε, Συμφωνία των Δημοσίων Αγορών και Προμηθειών. Γι' αυτό περιλαμβάνω αυτή τη μνήμα της Κίνας. Βεβαίω υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί στρατηγικοί εταίροι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, με τους οποίους έχουμε κρεμεί θέματα και ιδίω σε ό,τι αφορά την κάποια ε, τσιγκουνιά θα έλεγα με την οποία ανοίγουν τις αγορές τους οι χώρες αυτές. Θα τα συζητήσω αυτά με τους σκιώδεις. Βεβαίω και για τις επενδύσεις. Συμφωνώ ότι η λέξη επενδύσεις δεν αναφέρεται τόσο πολύ μέσα στο κείμενο, αλλά όπως είπα αναμένω και τις τροπολογίες σας. Δεν ήθελα να σας υποβάλω ένα κείμενο ήδη ολοκληρωμένο, κλειδωμένο εντό εισαγωγικών. Θα ενταχθεί βεβαίω και η πτυχή των επενδύσεων, αφού άλλωστε μιλούμε για αγορές και επενδύσεις ε, στη βάση προτάσεως που υποβάλλει η Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, εσείς θίξατε την αναγκαιότητα να υπάρξει περισσότερη συνοχή στις τεχνικές προδιαγραφές. Υπάρχει και μια παράγραφος συμπληρωματική που θα υπάρξει μάλλον, που μπορεί να περιλάβει τα θέματα αυτά, βεβαίως που είναι πολύ σημαντικά. Το ίδιο σχετικά με τα τελωνία, όντως εγώ δεν αναφέρθηκα διόλου στον ρόλο των τελωνίων και της τελωνιακής πολιτικής. Όπως είπα, δεν ήθελα να μπω και πολύ στα οικόπεδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θεώρησα ότι για την ώρα αυτά ήταν τα θέματα στα οποία θα ενέκυπτε η, έχει εγκύψει ήδη μάλλον η Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτού. Βεβαίως, είμαι διατεθειμένη να περιλάβω και την διάσταση αυτή που δικαίως τονίσατε. Θα ζητήσω συγγνώμη αν δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Το ζήτημα τώρα της ε, αεφόρου αναπτύξεως, όταν μιλούμε για αμοιβαιότητα στις συναλλαγές, αυτό γίνεται σε ένα πνεύμα σεβασμού των προδιαγραφών και στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οι εταίροι μας θα έλεγα ότι δεν σέβονται με την ίδια ας πούμε προσοχή και ένταση. Θα τονίσω λοιπόν και πάλι την ανάγκη τήρησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Όπως είπα, ζητώ συγγνώμη αν δεν απίτησα σε όλες τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις. Όπως είπα, ο διάλογος θα συνεχιστεί. Η ώρα περνάει. Θα περιοριστώ σε αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους για τις ε, παρεμβάσεις σας. Και όπως είπα θα προσπαθήσω να εντάξω όλες αυτές τις προτάσεις και τα σχόλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κείμενό μου, φροντίζοντας ταυτόχρονα να ρίξουμε το ιδιαίτερο βάρος στα θέματα αρμοδιότητας της ΕΜΚΟ της Επιτροπής μας δηλαδή, αλλά και την ευρύτερη ενατένιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι σημαντικός πλέον ισότιμος εταίρος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέος ρόλος αυτός για την Ευρωβουλή και ασφαλώς θα πρέπει να τον ε, παίξει σωστά. Well, thank you very much for that. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε από τις εκθέσεις, ε, από τις νομοδοτήσεις μας, υπάρχει περιορισμός ως ε, προς το, το μέγεθος της έκθεσης Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 12 έχουμε χρόνο για να προετοιμάσουμε τις τροπολογίες που θα σας αποστείλουμε και θα ψηφίσουμε στις 6 ε, Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ βραχή χρονοδιάγραμμα αλλά πρόκειται για μια ετήσια εκθέση όπως γνωρίζετε, άρα δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης. Δεν χρειάζεται να χρονοτριβούμε, άρα αναμένουμε τη συνεργασία μας μέχρι τότε. Άρα Φτάνουμε σε μία νέα έκθεση, τελευταία έκθεση για σήμερα το πρωί, που αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό. Άρα, καλώ την πρώτη αντιπρόεδρο, την κυρία Κορχόλα, να μας εισηγηθεί αυτή την έκθεση, η οποία, αυτή τη γνωμοδότηση, και μετά έχουμε τους Τα Ταραμπέλα από τους ασελστές Μάντερς ο κύριος Μάντερς μπορεί να εμφανιστεί τους πρασίνους. Η κυρία Μακλάρκιν έφυγε για μία συνέντευξη, ραδιοφωνική συνέντευξη, άρα θα αντικατασταθεί. Ε, υπάρχει και το θέμα των, ε, των τυχερών παιχνιδιών, το οποίο θα μας απασχολήσει αργότερα. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας, άρα δίνω το λόγο στην κυρία Κόρχολα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αρκετές ε, πτυχές. Ε, μιλάμε για την καταπολέμηση του ντοπαρίσματος, ε, ελεύθερη μετακίνηση αθλητών, διεθνή συνεργασία, εμείς θα ασχοληθούμε με την οικονομική διάσταση. Μιλάμε δηλαδή για τα τυχερά παιχνίδια, για τα στοιχήματα, πνευματικά δικαιώματα και την πώληση, διακρατική πώληση ε, εισιτηρίων. Όπως ξέρετε υπάρχουν πολλές οικονομικές επιπτώσεις και με τις τρεις πρώτες παραγράφους ήθελα να σταθώ στην ε, συνεχή χρηματοδότηση του αθλητισμού από τον ε, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ε, μιλήσαμε και για τα θέματα αλληλεγγύης που αφορούν τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ φτωχών και πλουσίων. μιλάμε ιδιαίτερα για την χρηματοδότηση αυτή ευρέως φάσματος και νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να προωθούν τα αποκλειστικά δικαιώματα έτσι ώστε να, προ, να προστατεύουμε τον τομέα από, την παράνομη, από τον παράνομο ανταγωνισμό. Μιλάμε λοιπόν για τα βασικά αθλητικά τις βασικές αθλητικές δραστηριότητες και τις χρηματοοικονομικές πολιτικές. Η παράγραφος 4 αναφέρεται στην πνευματική διαδικασία, στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσα στα πλαίσια της εμπορικής εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή κατανομή εσόδων. Η παράγραφος αναφέρεται στην διάταξη της οδηγίας υπηρεσιών που απαγορεύει τις διακρίσεις γιατί πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι οι πωλήσει εισιτηρίων ε, online είναι πολύ πιο ε, ακριβή έφνη στην Ολλανδία παρά στην Ισπανία. Αυτή η οδηγία περί ε, δεν έχει εφαρμοστεί ενιαία και ικανοποιητικά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένω τα σχόλια και τις τροπολογίες σας μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ, Ρίτα. Ακούσουμε τους δυο Καλώς ε, Καλωσορίζω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι αρμόδιος για αυτό το θέμα, και θα τον καλέσω να ε, μιλήσει με τα, τους βουλευτές. Λοιπόν, ο κύριος Ταραμπέλα πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κόρχολα για το σχέδιο γνωμοδότηση. Συμφωνώ με όλους τι παραγράφου και καλά έκανε και επέμεινε σε όλα τα σημεία. Έχω να σα πω τα εξή πέντε συνοπτικά. Πρώτον, για τον αθλητισμό έχουμε πολλά να πούμε και βεβαίω θα περιοριστούμε στις δικές μας αρμοδιότητες Επιτροπή ΣΥΜΚΟ. Θέλω να τονίσω ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Ε, θα συζητήσουμε και στην έκθεση του συναδέλφου ε, Κρόιτσμαν. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχουν τα εθνικά λαχεία, ε, τα κρατικά λαχεία, τα δημόσια που επενδύουν σε όλα τα αθλήματα, προσπαθούν τουλάχιστον, όχι μόνο στο πρωταθλητισμό ή στα της ελίτ, αλλά και στα λαϊκά αθλήματα. Εδώ το BetClick, click, το big win, τα στοιχήματα ε, online. Εγώ είμαι λίγο οπαδός της West Ham ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπω η φανέλα να γράφει Betwin, βεβαίω, γιατί βγάζουν πολλά λεφτά, αλλά εδρεύουν στη Μάλτα ή στο Γιβραλτάρ, όπου είναι πιο ευνοϊκό το φορολογικό καθεστώ. Δεν ξέρω αν αυτέ οι ιδιωτικέ εταιρείε επενδύουν στο μαζικό αθλητισμό, μάλλον επενδύουν ε, στη μεγιστοποίηση του κέρδου του. Και αυτό είναι το κινητρό του και ο λόγο ύπαρξη. Ε, σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με τα κρατικά ε, ε, συστήματα στοιχημάτων και ελαχεία. Θέλω να ε, αναφερθώ στα εμπορεύματα, φανέλες ποδοσφαίρου και άλλα, θα μπορούσαν να ε, παράγονται στην Ευρώπη. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να επιβεύουμε, αλλά βλέπω τις φανέλες. Εγώ είμαι, ξέρετε, φανατικός του ποδοσφαίρου. Κάθε φορά αλλάζουν οι φανέλες, ε, γιατί αλλάζει ο σπόνσορας ή αλλάζουν οι, οι ρίγες στην Ιταλία, ας πούμε, εγώ είμαι παδός μιας ομάδας ε, ε, με ρίγες μαύρες και μπλε και κάθε χρόνο αλλάζει το φάρδος για να αλλάζει φανέλα. Πιο μικρές ρίγες, πιο φαρδιές ρίγες, εντάξει, ωραία. Ε, αυτό αφορά τι εταιρείε βέβαια παραγωγή αθλητικών ειδών, αλλά ίσω ξέρω εγώ δεν χρειάζεται να αλλάζουν κάθε χρόνο τι ρίγε. Τρίτον, υποστηρίζω και πάλι την κυρία Κόρχολα όταν μιλάει για την ανάγκη να καλυφθεί το έλλειμμα ανάμεσα στα πλούσια και στα φτωχά αθλήματα. Τι εννοεί τα ε, αθλήματα που ε, προσελκύουν τα μέσα ενημέρωσης και έχει και ένα σύστημα αλληλεγγύης που προτείνει βεβαίως πολλοί πρωταθλητές. Ε, ανάλογα με το άθλημά τους δεν μπορούν να ζήσουν από το άθλημα αυτό, αλλά πρέπει να έχουν και επάγγελμα. Ενώ κάποιοι άλλοι κατακλείζονται από τα χρήματα που κερδίζουν από τον αθλητισμό. Τέταρτον, ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών του αθλητισμού και των πολλών εθελοντών. Ε, οι εθελοντές πιστοποιούνται, θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη αυτή η αναγνώριση για να μπορούν να ασκούν και επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται. Από ό,τι φαίνεται για το ποδόσφαιρο γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά για την κολύμβηση όχι. Κάποιο που είναι προπονητή κολύμβηση στη Γαλλία δεν μπορεί να έρθει στο Βέλγιο να εργαστεί. Αυτό δεν είναι το άκρο Πέμπτον, σε όλα τα αθλήματα βεβαίω η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών θα πρέπει να είναι δεδομένη στα πλαίσια της ισχύουσα νομολογίας, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Οι μεταγραφές ε, των παικτών τραβούν την προσοχή μας μέχρι αύριο <laughs> που λύγει η περίοδος, γιατί είναι τεράστια, τρελά τα ποσά, πραγματικά εξωφρενικά. Και εδώ υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητάει συνολική ε, αναθεώρηση των μεταγραφών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θυμάστε πριν από λίγα χρόνια την απόφαση Μπόσμαν, περιβόητη στο ποδόσφαιρο, αλλά ποτέ ίσως δεν μετρήσαμε ε, την επίπτωση. Βεβαίως θετική για τους παίκτες, ε, ελευθερώθηκαν από αυτή την απόφαση, πλούτησαν κιόλα γιατί είναι πιο ανεξάρτητοι από τις ομάδες τους, αλλά τι γίνεται με στις ακαδημίες παικτών, τα φυτόρια παικτών, τα σχολεία στις ομάδες. Οι επενδύσεις δεν είναι σίγουρες γιατί η ομάδα δεν είναι πλέον ο κύριος, ε, δεν έχει το τελευταίο λόγο για τον παίκτη όπως είχε στο παρελθόν και αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε υπό τη πτυχή αυτή και το πρίσμα και τέλος. Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω κάτι που έγινε στη Λιέγη. Συνάντησα τον κύριο Πάουερς που είναι ε, πολύ γνωστός γράφο. Φεύγει από την RTBF, την κρατική τηλεόραση και πάει στην RTL, την ιδιωτική. Και μου συνέστησε ένα κύριο και ήταν ο Ζαν Μαρκ Μποσμάν που έφερε όλη αυτή την απόφαση Μποσμαν στο δικαστήριο. Και είναι διάσημη αυτή η υπόθεση όχι μόνο στο Βέλγιο, στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο όλο. Ε, και ο κύριος Μπόσμαν λοιπόν που ήταν ο αίτιος αυτή τη υπόθεση και έκανε διάσημο το δικηγόρο του που τρέχουν όλοι να το ρωτήσουν. Αυτό που έκανε δισεκατομμυριούχου ε, του παίκτε στην Ευρώπη είναι πανφτωχό. Γιατί μετά δεν τον έπαιρνε καμία ομάδα και παίρνει κοινωνικά επιδόματα ε, από το Δήμο του που μένει κοντά στη Λιέγη και σε λίγο θα αφιερωθεί και ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ στην υπόθεση του. Παράδοξο δεν είναι, βλέπετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και θυμίζοντας και το θέμα της απόφασης Μπόσμαν και πόσο σημαντικό είναι και χαίρομαι που είστε τόσο ενθουσιώδης ε, φίλαθλος. Αποουσιάζει ο κύριος Μάντερς, αλλά έχουμε άλλο μεγάλο οπαδό, τον κύριο Κρόιτσμαν. Τώρα μπορείτε να μας διαβάσετε και το δικό του ενθουσιασμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να συζητήσουμε κι εμείς για τα στοιχήματα στο διαδίκτυο, ε, είναι θέματα αδειών, είναι θέματα αθλητικών διοργανώσεων, αλλά κοιτάξτε εκεί ε, πρέπει λίγο να προσέξουμε και την αρχή της επικουρικότητας και να το συζητήσουμε βεβαίως, διότι αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη, όταν παίρνουν περισσότερα χρήματα από τα στοιχήματα στο διαδίκτυο, είναι δική τους υπόθεση, γιατί διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας. Πολλά κράτη βεβαίως ενισχύουν τον αθλητισμό, είναι σαφές. Αν κοιτάξετε καν η δική μου χώρα, ρέουν τα κονδύλια εκεί από το τολότο, το αντίστοιχο προπό και δεν είναι μόνο ε, υπέρ των ε, επαγγελματιών αλλά και υπέρ των αριστεχνών και ε, τον αθλητισμό γενικότερα. Διάβασα τη γνωμοδότηση. Δεν είναι σε μεγάλη αντίθεση με αυτά που συζητούμε στη δική μου έκθεση. Είναι πάνω από 200 οι τροπολογίες, αλλά τι γίνεται με την πνευματική ιδιοκτησία, είναι πάγιο θέμα. Πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συμπεριλάβουν και τα πνευματικά δικαιώματα εκεί. Ας το κοιτάξουν τα κράτη-μέλη αυτό μεταξύ τους, εάν θα έχουν μερίδιο στα κέρδη και οι διοργανωτές Αυτά. Κατά τα άλλα συμφωνούμε γενικά με την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Η κυρία Ρούλε, όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει να μιλήσει η κυρία Ρούλε. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος της ε, Μαρκ που είναι σκιώδης εισηγήτρια εξ ονόματος της ομάδας μας ε, μου ζήτησε να κάνω μερικά σχόλια. Πρώτον, να ευχαριστήσω την κυρία Κόρχολα για το σχέδιο γνωμοδότησης. Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αθλητισμό ε, απορρέουν από το άρθρο 165 της συνθήκης και αφορούν τον αθλητισμό ε, σε εθελοντική βάση και πραγματικά τον ερασιτεχνιστικό και δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό αθλητισμό ελίτ. Η κυρία Μακλάρκιν ε, θεωρεί ότι τα στοιχήματα συνεισφέρουν σημαντικά στη χρηματοδότηση του αθλητισμού. Ε, δεν θεωρεί ότι η παράγραφος 3 είναι πρακτική λύση για να ε, προστατευτούν κάποιες εταιρείε. Επίσης, γίνεται μια διάξη ανάμεσα σε πλούσια εντός εισαγωγικών και φτωχά εντό εισαγωγικών αθλήματα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η χρηματοδοτική αλληλεγγύη και ο αντίστοιχος μηχανισμός είναι ε, δίκαιο μέσο και εργαλείο για όλα τα αθλήματα και σας ρωτώ και ποιο παρακαλώ θα ε, αποφασίζει ποιο άθλημα είναι πλούσιο και ποιο είναι φτωχό και ποιο θα αποφασίσει πώς θα μοιραστούν τα χρήματα και στη συνέχεια τι θα γίνει, τι άλλο θα δούμε. Ένα ευρωπαϊκό ταμείο ή φορέα ή agency για την αλληλεγγύη στον αθλητισμό και να βασιστεί να έχει και έδρα μάλλον κάπου μακριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολύ μεγάλο οργανόγραμμα, με παχυλούς μισθούς και ακόμα παχυλότερες συντάξεις για τους υπαλλήλους. Και αν μπορώ να πω κάτι στον κύριο Ταραμπέλα, άκουσα αυτά που είπατε για τα προβλήματα ε, με τις φανέλες και τις ομάδες που κάθε μήνα έχουν ε, άλλα ε, εξαρτήματα άλλες Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο. Και δεν θα πούμε εμείς τις ομάδες κάθε πώς θα αλλάζουν φανέλα και με ε, τι ρυθμό. Μπορεί να σας φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθεί παρά να ανακατεύεται σε τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε στα μεγάλα και σημαντικά θέματα. Η κυρία Μακλάκιν δεν πιστεύει ότι η πώληση των εισιτήριων για αθλητικές διοργανώσεις θα πρέπει να ε, εμπίπτει στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Βλέπουμε ευνοϊκά και κατανοούμε την πρόταση της εισηγήτριας, αλλά θα ήταν πάρα πολύ ζήμιο αυτό για τις μικρές ε, ομάδες, τους μικρούς συλλόγους και σωματεία που πολλούν με αυτόν τον τρόπο εισιτήρια στους φιλάθλους. Ε, ευχαριστούμε και θα κάνουμε και τις τροπολογίες μας, λέει η κυρία Μακλάφιν. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάλτε Μόζε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εντάχει να πω ότι πρόκειται για, μια, για ένα πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης και στο σημείο Α αναφέρεται ότι θα πρέπει να, δούμε, να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική πτυχή του αθλητισμού καθώς και θέματα ε, υγείας έχουν μεγάλη σημασία για τα βασικά αθλήματα. Όταν μιλάμε για την αρχή της επικουρικότητας και για τη, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια, ε, δέχομαι την διατύπωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι δεν μιλώ ως μέλος ε, της ΙΜΚΟ, αλλά της Γεωργικής Επιτροπής. Δεν θα ήθελα να λάβω υπόψη τις μεμονωμένες προτάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κορχόλα. Συμφωνώ με την ε, κυρία Σαλτεμόζερ ότι θα πρέπει να δούμε θέματα υγείας και έχουν διενεργηθεί μελέτες που καταδεικνύουν ότι ο αθλητισμός έχει μεγάλη σημασία για τον τομέα της υγείας. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή, ίσως όχι τώρα, αλλά να ε, ασχοληθεί με θέματα αθλητισμού στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 γιατί υπάρχουν ε, ε, μέλη του Κοινοβουλίου που θέλουν να υποβαθμίσουν τον αθλητισμό και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να το δεχτούμε, διότι είναι ένα θέμα ύψης της ε, πολιτικής σημασίας και θα πρέπει να προωθήσουμε την στρατηγική 2020. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή αυτή να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα του αθλητισμού. Άλλοι που θα ήθελε να συνεισφέρουν φαίνεται πως όχι. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ο κύριος Βελάφκεθ. Ίσως θα μπορούσε να λάβει το λόγο και μετά η κυρία Κορχόλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να παρέμβω εδώ. Όπως ε, είπατε, είμαι υπεύθυνο της ε, υπηρεσίας αθλητισμού μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ασχολούμαστε με τις νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του αθλητισμού. Πρόκειται για το άρθρο 165 που ασχολείται με το συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών και δεν μπορεί να γίνει ε, πλήρης εναρμόνιση σε αυτό το τομέα. Μέσα στα πλαίσια της ανακοίνωσης που ασχολείται με την ανάπτυξη του αθλητισμού, στην ανακοίνωση αυτή προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό σε όλες τις διαστάσεις του μέσα στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων. Μία από τις ε, δυσκολίες που καταδεικνύει αυτή τη δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στον αθλητισμό να ξεχωρίσουμε τη μία πτυχή του από άλλες δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τον αθλητισμό της ελίτ ή με τον φτωχό αθλητισμό. Αυτό που ονομάζεται grassroots sport. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ο επαγγελματικός αθλητισμός επηρεάζει και τον φτωχό αθλητισμό και να δούμε κατά πόσο αυτά τα μέτρα της ε, Κομισιόν που προβάλλονται ε, μέσα στα πλαίσια το 165 προβάλλουν και άλλα μέτρα ρύθμισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε άλλους τομείς που δεν έχουν σχέση άμεσα με τον αθλητισμό αλλά σχετίζονται με τον τρόπο ρύθμισης ή χρηματοδότησης του αθλητισμού. Το είδαμε με την οδηγία περί υπηρεσιών, περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, περί ανταγωνισμού, περί αθλητισμού, χρηματοδότησης του αθλητισμού και θέματα λαχιοφόρων αγορών στα πλαίσια του αθλητισμού. Αυτά εν είδη εισήγησης θα ήθελα να πω ότι αυτά τα στοιχεία που εντάσσονται στο σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής σας. Αυτά τα στοιχεία θα αναθεωρούν θέματα που έχουν ρυθμιστεί στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Και αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ όπως το θέμα της ε, χρηματοδότησης του βασικού λαϊκού αθλητισμού είναι θέματα που απασχόλησαν και αυτή τη μελέτη ή αυτές τις μελέτες που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν και θα ασχοληθούμε με τον βασικό λαϊκό αθλητισμό και στις μελλοντικές μελέτες ως προς τους μηχανισμούς αλληλεγγύης που προβάλλονται εδώ η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εμείς επιμείναμε σε αυτή την πτυχή στην ανακοίνωση, δηλαδή ότι χρειάζεται ε, αλληλεγγύη μεταξύ επαγγελματικού και μη αθλητισμού. Αυτό το λένε και οι μεγάλοι ε, επαγγελματικοί ε, όμιλοι, η UEFA, η FIFA, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και ούτω καθεξής. Πρόκειται για μηχανισμούς αλληλεγγύης που χρειάζονται έτσι ώστε η βασική αυτή χρηματοδότηση που προκύπτει από τον επαγγελματικό αθλητισμό να χρηματοδοτεί τον λαϊκό αθλητισμό. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η αλληλεγγύη, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε και όπως τονίσατε και στην ανακοίνωση θα πρέπει να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε αυτούς τους μηχανισμούς αλληλεγγύης. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, την προστασία των ταμείων ή των χρωματοδοτήσεων μέσω λαχιοφόρων αγορών και αυτές τις χρηματοοικονομικές εισρωές για τον λαϊκό αθλητισμό. Ως προς το θέμα που τίθεται για τα τυχερά παιχνίδια online και τα στοιχήματα, ξέρετε ότι πρόκειται για μια παράλληλη διαδικασία για τα στοιχήματα online. Αυτή τη στιγμή συντάσσεται μία πράσινη βίβλος και πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία της Κομισιόν θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω σκέψεις και εξελίξεις και θέλουμε και τη δική σας γνωμοδότηση. Ως προς τα θέματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία προαναφερθήκατε, προαναφέρθηκα και εγώ, και ως προς την πώληση εισιτηρίων, ως προς, ως προς το σημείο 5, θα ήθελα να πω ότι δεν καλύπτεται ιδιαίτερα στην ανακοίνωσή μας, αλλά εφόσον το θέσατε εσείς και εμείς θα το παρακολουθήσουμε για να δούμε πώς ε, εξελίσσεται το θέμα των διασυνοριακών πωλήσεων. μέσα στα πλαίσια της δικής σας εισήγησης. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ για την εκτενή σας παρουσίαση και γιατί μας ε, υπενθυμίσατε για ορισμένες νέες αρμοδιότητες Επιτροπής Δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η κυρία Κορχόλα, θέλετε το λόγο για να συνοψίσετε και να μας επιβεβαιώσετε το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σκόπιμα αυτά σχόλια. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξισορροπημένη προσέγγιση Ευχαριστώ και την Επιτροπή μας εξηγήσατε γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε, να ασχοληθούμε και με τα φτωχά αθλήματα και να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών αθλημάτων. Βεβαίως τα θέματα της υγείας δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ όταν μιλάμε για αθλητισμό. Αυτή η έκθεση όμως ήταν έκθεση της ΙΜΚΟ και γι' αυτό ασχοληθήκαμε με την οικονομική διάσταση ε, στρίκτο σένσου. Βεβαίως υπό την ευρύτερη έννοια θα έπρεπε κανείς να ασχοληθεί και με την υγεία και την οικονομική διάσταση της υγείας. Χρονοδιάγραμμα τώρα. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 2 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί. 19 Σεπτεμβρίου για να εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ την ίδια ημέρα, στις 19 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Στην Επιτροπή Πολιτισμού θα γίνει ψηφοφορία κατά τις αρχές Οκτωβρίου. 4-5 Οκτωβρίου σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Υπάρχουν, νομίζω θα υπάρξουν ε, πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Σήμερα το πρωί λυπάμαι διότι είχαμε μία αργή εκκίνηση και δύσκολη εκκίνηση λόγω τεχνολογικών προβλημάτων. Θα συναντηθούμε στις 3 το απόγευμα και θα ασχοληθούμε με δύο βασικές εκθέσεις θέσεις. Ε, θα μιλήσουμε για τα γεωργικά και δασικά οχήματα και για τις αγορές δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων. Θα τα πούμε στις 3. Ευχαριστώ.